Καθίστε τώρα. Καλημέρα. Είναι κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης Εξωτερικών Υποθέσεων των δύο επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη. Το ένα είναι η έγκριση ημερήσιας διάταξης δεν με ειδοποίησαν οι αλλαγέ αυτή. Υποθέτω ότι εγκρίνεται το σημείο 1. Σημείο 2. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Δεν υπάρχουν ανακοινώσει. Σα ευχαριστώ. Συνάδελφοι, τώρα θα πάμε στο βασικό σημείο της έκτακτης αυτής κοινή συνεδρίασης της έναρξης του νέου προγράμματος «Ανταπόκριση στα προβλήματα του Ιράκ». Είναι σημαντικότατη αυτή η διάσκεψη και εκ μέρους των Επιτροπών Ανάπτυξη Εξωτερικών Υποθέσεων θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά όλους σα εδώ σε αυτή την ε, συνεδρίαση υψηλό επίπεδου που συνοργανώνεται ε, μεταξύ, συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Ηνωμένων Εθνών και ε, συμμετέχουν οι Επιτροπές Εξωτερικών και ανάπτυξη Λοιπόν, είναι πολύ επίκαιρη στιγμή που συζητάμε αυτό το θέμα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και υποχρέωσε σχεδόν 3 εκατομμύρια ανθρώπου να φύγουν από τα σπίτια του. Άφησε πάνω από 8,2 εκατομμύρια ανθρώπου που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτά τα στοιχεία είναι ε, εκπληκτικά μα καταθλίβουν και υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Περνάνε τα πάνδυνα. Ε, λοιπόν, εμποδίζει, εμποδίζουν η βιοπραγία στη χορήγηση βοήθειας και ε, κλιμακώνεται η σύραξη και γίνονται φοβερές βιοπραγίες από το ISIL και οπότε πρέπει να προστατευτούν οι ευάλωτες ε, ομάδες, κυρίως οι γυναίκες και τα παιδιά και είναι κατεπίγουσα αυτή η ανάγκη. τα, περισσότερα παιδιά πρόσφυγες και τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στην παιδεία και η παιδική του ηλικία σημαδεύεται από σύγκρουση, βιοπραγία και υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν ψυχικά και φυσικά βέβαια Έχουμε τι ευρωπαϊκέ ημερίδε ανάπτυξη. Χθε που μιλούσα σε μια εκδήλωση, σε διάφορου χρηματούχου μου έλεγαν ότι κατά μέσο όρο οι εκτοπιστέντε, ε, ομοιέ ηλικία έχουν μείνει 17 χρόνια εκτοπιστέντες ε, μεγάλο χρονικό διάστημα όλη η παιδική σου ηλικία και η εφηβεία σου περνά χωρίς την ε, εκπαίδευση και αυτό είναι κατεπήγον θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα στο Ιράκ και να αντιμετωπιστούν οι ανθρωπιστικές ε, ανάγκες και θα πρέπει να εστιαστούμε επί της παιδείας για αυτή την γενιά. Λοιπόν, τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μένα σήμερα το πρωί που καλώς ορίζω την κυρία Κιούμγα Καν που αναπληρώνω ότι έγινε και ε, Γραμματέα για τα Ανθρωπιστικά Θέματα και Συντονίστρια για την Βοήθεια που παρέχει ο ΙΕ και κύριο, τον κύριο Χρήστο Σιλιανίδη που είναι επίτροπο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση των Κρίσεων. Η κυρία Καν, είναι τιμή μα που είσαστε εδώ, αντιπροσωπεύετε τον ΟΗΕ και το εστιακό σημείο που αφορά τι καταστροφέ και την υπηρεσία συντονισμού των ανθρωπιστικών ε, ενισχύσεων και που προσπαθεί να συντονίσει τη διασωσφάση που καταβάλλονται και τη χρηματοδότηση για ανθρωπιστικού σκοπού. Ε, Πίτροπε κύριε Στυλιανίδη, είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε ξανά εδώ ε, οι Επιτροπέ Ανάπτυξη και Άφετη καταστρώσαν τη στρατηγική τη σηματοδοσία του Ιράκ για τη Συρία τη Ευρωπαϊκή Ενώσει που έχουν καταστραφεί από αυτή την παρατεταμένη σύγκρουση, σύραξη. καλούμε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια και σε εκείνου που πλήττονται στο Ιράκ. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να δράσουμε μαζί ούτω ώστε η χρηματοδότηση να διατεθεί, η απαιτούμενη. Κύριε Μπροκ, ε, θέλετε να πείτε κάτι, μερικά λόγια. Αν μου επιτρέπετε, λέει ο κύριος Μπρόκ. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς, ο κύριος Μπρόκ. Χωρίς μικρόφωνο, ο κύριος Μπρόκ. debate σας ευχαριστώ. Ε, η σημερινή μας συνεδρίαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, μόλις ζητούσαμε τον πρόεδρο του Ιρακινού Κοινοβουλίου και πρέπει να πω ότι είναι τεράστια σημασία η κατάσταση και θα πρέπει να δημιουργηθεί μια σταθερότητα. Αύριο θα ηγηθώ μια αντιπροσωπεία ε, που θα μεταβεί στην Τεχεράνη και όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να ειδωθούν από κοινού σε ένα συνολικό πλαίσιο έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Αν δεν μπορέσουμε να το καταφέρουμε σε μια χώρα σαν το Ιράκ, αν δεν υπάρξει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ε, να συμμετέχουν όλα τα τμήματα της κοινωνίας, θα έχουμε τεράστια προβλήματα γενικότερα Εάν η σουνητική μειονότητα της χώρας δεν έχει την αίσθηση ότι είναι ισότιμος εταίρος και έχει ρόλο να διαδραματίσει, τότε θα είναι δύσκολο να βρεθεί αξιοπιστία για να καταπολεμηθεί το Ισλαμικό κράτος. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που συζητούμε και θέματα ανθρωπιστικά αλλά και ε, αναπτυξιακά του Ιράκ, αλλά θα πρέπει να υπάρξει πρώτα σταθερότητα και η σταθερότητα να εδράζεται ε, σε οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους. Αυτά είναι κομβική σημασία ζητήματα. Επίσης, χαιρόμαστε για την παρουσία της ε, αναπληρώτριας Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και ε, του δικού μας Επιτρόπου. Χαίρομαι που ήρθαν να μας εξηγήσουν τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Επίσης, ε, χαιρόμαστε πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τον πρόεδρο της Ιρακινής Βουλής και με άλλους. Και χαίρομαι που ξαναβλέπω τον παλιό μου φίλο Τόνι Λέικ. Από προηγούμενες ιδιότητες είχαμε συναντήθει στη ζωή μας. Ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα έχουμε, ελπίζω, μια γόνιμη συζήτηση για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ό,τι μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εύχομαι να γίνει καλή συζήτηση. Ε, ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στους βασικούς μας ομιλητές για σήμερα το πρωί. Θα δώσουμε το λόγο πρώτα στην κυρία ε, Καν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Μπρόκ, Επίτροπε κύριε Στυλιανίδη, εξοχότητές σας κυρία Αλτζαμπούδη και διακεκριμένα μέλη της Ιρακινής Αντιπροσωπείας εξοχότητες κυρίες και κύριοι εκ μέρους ε, του ΟΗΕ, του Γενικού Γραμματέα του κ. Μπάνκιμεν και του νέου συντονιστού του κ. Στίβεν Ομπράιν για τις κατεπίγουσες ανάγκες και όλων των εταίρων που προσπαθούν στο Ιράκ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά που είσαστε εδώ παρόντες για να δείξετε αλληλεγγύη στο λαό του Ιράκ Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φιλοξενεί αυτή την εκδήλωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΚΟ και τους λαούς της Ευρώπης διότι ηγείστε στις ανθρωπιστικές δράσεις στο Ιράκ και σε όλο τον κόσμο. Εξοχότητες, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία, τους τελευταίους 18 μήνες ο λαός του Ιράκ έχει υποφέρει μια φρικτή τραγωδία η οποία συνεχίζεται να εκτιλήσεται και σήμερα. Πριν από ένα χρόνο περίπου μισό εκατομμύριο Ιρακινοί έπρεπε να το σκάσουν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, λόγω αυξανόμενων αβιοπραγιών στο Άνμπαρ μεταξύ ε, του Ιρακινού κράτους ε, και άλλων ομάδων και της Ιρακινής κυβερνήσεως. Διπλασιάστηκε ο αριθμός τους διότι μεγάλα ποσοστά της χώρας μπήκαν στον έλεγχο του Ισλαμικού κράτους. Σήμερα περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό τη χώρα. Πολλέ οικογένειε έπρεπε να μετακινηθούν πολλέ φορέ, ούτω ώστε να προηγούνται κατά ένα βήμα από τι φρικτέ βιοπραγίε, οι οποίε σαρώνουν ολόκληρε περιοχέ τη χώρα. Άλλοι δεν γνωρίζουν πού μπορούν να βρουν την ασφάλεια διότι έχουν παγιδευτεί σε μια διαίρεση ε, των διαφόρων ομάδων και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Κάθε ένας από αυτούς τους, τα τρία εκατομμύρια ανθρώπους είναι ένα παιδί, μια γυναίκα, ένας άντρας που έχουν υποχρεωθεί να φύγουν από ένα γνωστό περιβάλλον για να ξεφύγουν προς αβέβαιο μέλλον. Πρόσφατα 237.000 άνθρωποι ξέφυγαν από το Ραμάντι όταν έπεφτε η ε, πόλη στον έλεγχο της ομικού κράτους. Πάνω από ένα εκατομμύριο Ιρακινοί χρειάζονται καταπήγουσα βοήθεια και προστασία. Όλα τα κομμάτια, οι ομάδες της Ιρακινής κοινωνίας, οι Εζίδοι, οι Χριστιανοί, οι Σαμπάκ, οι Τουρκμένοι, οι Σουνίτες, οι Σιήτες και οι Κούρδοι έχουν πληγεί από τις οπραγίες. Η οικονομία έχει ε, πληγεί και η γεωργική παραγωγή έχει μειωθεί. Τα νοσοκομεία και διάφορες μονάδες περίθαλψης έχουν υποστεί βλάβες και έχουν καταστραφεί εκατοντάδες σχολεία, έχουν χρησιμοποιηθεί σαν σημεία για κατεπίκους ανάγκες ή για στατιωτικούς σκοπούς, ακόμα και σε ασφαλείς περιοχές η ανεργία και το κόστος ε, της διαβίωσης έχουν αυξηθεί και τα, οι αμοιβέ έχουν ε, μειωθεί. Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν απαχθεί, έχουν υποστεί συστηματική σεξουαλική βία και σκλαβιά και δουλεία. Κάποια παιδιά έχουν υποφέρει την απώλεια των γονιών τους, άλλοι έχουν υποχρεωθεί να πολεμήσουν ή να, να το για να προστατεύσουν τη ζωή τους. Οι εκτοπιστέντες οι οικογένειες ε, προστατεύουν οπουδήποτε γίνεται ε, σε κτίρια, εγκαταλειμμένα κτίρια, στα δίπλα στους δρόμους, στο πλάι των δρόμων και σε διάφορα σημεία ελέγχου, ενώ περιμένουν να περάσουν ασφαλείς περιοχές. Δεν έχουν πρόσβαση στις πιο βασικές υπηρεσίες όπως είναι η στέγαση, πόσιμο καθαρό νερό, η περίθαλψη υγείας και η παιδεία. Κυρίες και κύριοι, σε ανταπόκριση σε αυτή την απελπιστική κατάσταση, ο ΙΕ και οι εταίροι του ΟΗΕ έχουν κλιμακώσει δραματικά τα προγράμματά τους εντός της χώρας το τελευταίο χρόνο. Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο Ιράκ τώρα είναι από τις μεγαλύτερες και περιπλοκότερες στον κόσμο και παρέχουν υποστήριξη σε πάνω από 2 εκατομμύρια Ιρακινούς σε κάθε ε, περιοχή της χώρας κάθε μήνα. Ε, τρόφιμα, εμφιαλωμένο νερό και βασικά ε, αντικείμενα που είναι απαιτούνται για την επιβίωση ε, διαβιβάζονται στον κόσμο, μοιράζονται στον κόσμο, στι άκρε των δρόμων και σε σημεία ελέγχου. Εκατομμύρια άνθρωποι ε, βοηθούνται καθημερινά ε, μέσω διαφόρων πακέτων διατροφή που σχορηγούνται και, και στι διάφορα νοσοκομεία κλπ. παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και γυναίκε που έχουν υποστεί ψυχολογικά τραύματα. Αυτά τα ανθρωπιστικά προγράμματα όμω απειλούνται σοβαρά λόγω ελλείψεω χρηματοδότηση. Χωρί περισσότερη υποστήριξη, περίπου 50% των ανθρωπιστικών προγραμμάτων μπορεί να περικοπούν ή να σταματήσουν να εφαρμόζονται ξεκινώντα ε, τι δύο επόμενε εβδομάδε. Υπάρχει ένα πραγματικό κίνδυνο εκατομμύρια άνθρωποι να μην έχουν καθαρό νερό, να μην έχουν τροφή ούτε να έχουν και τι βασικέ υπηρεσίε. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα να ξεκινήσουμε την ανθρωπιστική ανταπόκριση και το σχετικό σχέδιο ανταπόκριση για το Ιράκ που βασίζεται σε επικαιροποιημένη στρατηγική που αντικατοπτρίζει την επιδεινούμενη κατάσταση το τελευταίο εννέα μήνο. Το σχέδιο λοιπόν ζητά 497,9 εκατομμύρια δολάρια, ούτω ώστε να παρασχεθεί βοήθεια που θα σώσει ζωέ και προστασία να παρασχεθεί σε 5,6 εκατομμύρια ανθρώπου στο Ιράκ για το υπόλοιπο έτο. Όλη η ανθρωπιστική κοινότητα χρειάζεται την βιώσιμη βοήθειά σα, ούτω ώστε να εξακολουθούμε να στηρίζουμε του Ιρακινού που έχουν ανάγκη. Όλοι είδαμε αυτή την κρίση να εκτελήσεται με τον πλέον δραματικό τρόπο στι τηλεοπτικέ μα οθόνε και στι οθόνε των υπολογιστών μα από την βία κατάκτηση της Μοσούλης, τις εικόνες οικογενειών που είχαν απομονωθεί στο όρο Σιντζάρ και την πρόσφαση πτώση του Ραμάντι. Ο λαός του Ιράκ ζει αυτή την καταστροφή καθημερινά. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για να σταματήσει η βία. Όμως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους βοηθήσουμε. Ο λαός του Ιράκ χρειάζεται τη βοήθειά μας τώρα. Αυτό το σχέδιο ανθρωπιστική ανταπόκριση δίνει ένα συγκεκριμένο δρόμο που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις κατεπίγουσες ανάγκες των γυναικών, των κοριτσιών, των αγοριών και των ανδρών στο Ιράκ. Δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε αβοήθητους. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος Τηλιανίδης θα πάρει τώρα το λόγο. Αγαπητή Λίντα, αγαπητέ Έλμαρ. Πρέζει πρέσβης Αλτζαμπούρη Σίντι. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Αναπτυξιακών Ζητημάτων για τη διοργάνωση ε, της σημερινής συνάντησης Έλμαν Μπρόκ, Λίνα Μακέβαν. Σας ευχαριστώ έχετε καταδείξει επανειλημμένα τη δέσμευσή σας ε, για να βοηθήσετε ε, τους Ιρακινούς πολίτες να υπερβούν τις τραγικές συνέπειες ε, του πολέμου και να φτιάξετε ένα καλύτερο μέλλον για την επόμενη γενιά Ιρακινών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Δόκτωρ Σαλίμ Αλ Τζαμπούρη, τον πρόεδρο δηλαδή του Ιρακινού Κοινοβουλίου και τον Δ. Αλή Σίντι, Υπουργό εγωταξικού Σχεδιασμού της ε, κυβέρνησης ε, του Κουρδιστάν στο Ιράκ. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην ε, σημερινή εκδήλωση. Αγαπητοί φίλοι, έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο, ένας χρόνος από το πρώτο κύμα εσωτερικά εκτοπιστέντων και συνεχίζει η χώρα να υποφέρει από μια καταστροφική σύραξη που έχει δημιουργήσει μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις της σημερινής εποχής. Θα ήθελα με τη σημερινή ευκαιρία να εκφράσω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδικάζοντας τις τρομοκρατικές μεθόδους, τις καταστροφικές δράσεις του Ίζιλ. Θα επισκεφθώ σύντομα τη Βαγδάτη και ο στόχος της αποστολής μου είναι διτός. Πρώτον, θα ήθελα κατηδίαν να εκφράσω την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους πολίτες και προς την κυβέρνηση, να τους διαβεβαιώσω ότι είναι ισχυρή και μακροπρόθεσμη η δέσμευση που έχουμε αναλάβει και δεύτερον, θα ήθελα να διώσω η διεισόμαση την κατάσταση επιτόπου ώστε να αποτιμήσω την κατάσταση και να εντοπίσω ε, τα κενά. Θα επισκεφθώ καταβλισμούς εσωτερικά εκτοπιστέντων στη Βαγδάτη ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους ε, από διάφορες πόλεις και χωριά, από το Ραμάτι παραδείγματος χάρη, πάνω από 200.000 άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους. Θα είμαι εκεί στο πλευρό τους για να τους ακούσω, για να ακούσω τις τρομακτικές τους εμπειρίες, τις ανησυχίες που έχουν και να τους διαβεβαιώσω ότι δεν είναι μόνοι τους. Αναπληρωτρία Γενική γραμματέα. η κυρία Γκάγκ, μας έδωσε τις ε, τα τρομακτικά στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την ανθρωπιστική τραγωδία του Ιράκ. Πάνω από 8 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται απεγνωσμένα τη βοήθειά μας. Ε, σχεδόν ε, τα 4 εκατομμύρια είναι παιδιά. Έχει σημειωθεί 400% αύξηση σε αυτό το τρομακτικό είδη αριθμό τα, τα, τα τελευταία χρόνια. Έχει αντιτικοποιηθεί, κλιμακωθεί σύραξη σχεδόν 2 εκατομμύρια ακόμη θα εκτοπιστούν μέχρι το τέλος του 2015, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Αυτή η κρίση πλήττει ολόκληρη τη χώρα και όλες τις κοινότητες. Θα δούμε και ένα βίντεο τώρα στη συνέχεια που θα μας δείξει το πραγματικό πρόσωπο αυτής της τραγωδίας. Αυτοί οι άνθρωποι εξαρτώνται απολύτως από τη δική μας βοήθεια. Η ευθύνη είναι συλλογική για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Η αλληλεγγύη μας θα πρέπει να παραμείνει απτή. Επικροτώ ε, το ότι ε, ανταποκρίνεται στο ηθικό της καθήκον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την αρχή της κρίσης είμαστε από τους μεγαλύτερους δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας ε, στο Ιράκ. Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι στην πρώτη θέση και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη γενναιοδορία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στη δεύτερη θέση. Όμως θα πρέπει να επιδιώξουμε μια επίρρωση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, διότι η ανθρωπιστική ε, δράση στο Ιράκ ε, υποχρηματοδοτείται σε κρίσιμο σημείο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να αφήνουμε εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό, σε τροφή, σε στέγη, σε υγειονομική περίθαλψη. Τα βασικά δηλαδή που χρειάζεται κανείς για να επιβιώσει είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Πέραν αυτού, η κατάσταση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη απειλή για την ασφάλειά μας, διότι αποσταθεροποιεί ολόκληρη τη χώρα αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Τροφοδοτεί το φαύλο κύκλο της βίας και του κατακαιρματισμού. Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης προσαρρογή των ε, θυμάτων της κρίσης δεν συνιστά μόνο ένα ηθικό καθήκον. Είναι μια επιτακτική ανάγκη για λόγους ασφάλειας και γι' αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί σε ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις Ιρακινές Αρχές, για την διεθνή κοινότητα. Η υποστήριξη που προσφέρουμε θα πρέπει να υπακούει σε βασικές αρχές. Θα πρέπει να είναι καθολική, ε, και διαθέσιμη σε όλους τους ευάλωτους, να βασιζόμαστε σε ανάγκες και όχι σε ε, μικροκομματικές σκοπιμότητες, σεβόμενοι την θρησκευτική διαφορετικότητα, τις διάφορες κοινότητες που υπάρχουν, καθώς και ε, μη λαμβάνοντας υπόψη τυχόν γεωγραφικές, ε, γεωγραφικού χαρακτήρα δυσκολίες για την πρόσβαση στα θύματα. Προτού αρχίσουμε τις συζητήσεις, ας ε, παρακολουθήσουμε το βίντεο του ΟΗΕ για την ε, επιτόπου ε, δράση της ομάδας που είναι αρμόδια για το Ιράκ. يعني هذا صار بعد ما يعني ما Μα Ένα Ιρακινό δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ρόλο να παίξει. Είναι μηδαμινό. Τι είναι αυτά. Υπό την απειλή των όπλων μας έκαναν να φύγουμε από τα σπίτια μας. Φύγαμε, κανείς δεν ήρθε να μας βοηθήσει. Στην περιοχή όπου ζούμε όλος ο κόσμος μας, μας μισεί. Στο Ιράκ μια ανθρωπιστική τραγωδία εξακολουθεί να εκτιλήσεται επιθέσεις από εξαμιστικές ομάδες έχουν διαδώσει τη βία στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Σαν αποτέλεσμα από τον Ιανουάριο του 2014 2,9 εκατομμύρια τρομοκρατημένοι πολίτες έχουν ξεφύγει από τις πόλεις τους. Προσπαθούν ε, να πάνε να στεγαστούν σε διάφορους καταβλισμούς. Οι εκτοπιστέντες έχουν γίνει μια τεράστια πρόκληση για το Ιράκ έχουμε κατεπηγόντως ανάγκη βοήθεια από τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και από άλλες ε, οργανώσεις ούτως ώστε να μας δώσουν βοήθεια και να μπορούμε να την ε, μοιράσουμε. Μετά το ξέσπασμα της κρίσης, οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες έχουν δώσει τρόφιμα, βοήθεια, νερό, γενομική περίθαλψη, κατεπίγουσα βοήθεια όσον αφορά τις διάφορες ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία, βοηθούν τον κόσμο να επιβιώσει, βοηθούν τα ευάλωτα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους, τους παρέχουν προστασία. Μετά την αρχή της κρίσης ε, έχουμε αυξήσει τον προπολογισμό, έχουμε ανοίξει τα σπίτια μας στους ανθρώπους αυτούς για να τους δώσουμε βοήθεια. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση μόνοι μας και επιπλέον είναι διεθνής ε, ευθύνη Ήρθα θα λέμε ότι πρέπει να μείνω εδώ για μία εβδομάδα, δύο εβδομάδε. Ε, δεν ξέρω πώ θα τα καταφέρω. Κάθε μέρα είναι δύσκολη. Έχω νέα παιδιά, ε, μικρά παιδάκια που είναι δίδυμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα φροντίσω εδώ πέρα. Πραγματικά δύσκολο να τα φροντίσω τα παιδιά. Προσπαθούμε να τα κατάμε δροσερά με νερό. Το τι έκανε αυτό το παιδάκι, σε τι φταίει το παιδάκι. Πρέπει να ζει σε ένα αντίσκηνο, στη μέση της ερήμου. Και όπω επιφυλάσσεται τώρα ένα καλοκαίρι γεμάτο συγκρούσεις, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί έτσι περαιτέρω. Οι υπηρεσίε ε, για εκατομμύρια από ευάλωτου ανθρώπου ε, που παρέχονται σε αυτού, εξαρτώνται ε, από βοήθεια και οι υπηρεσίε μένουν από χρήματα. Δεν έχουν μείνει χρήματα. Εντός, ενός, εντός μηνών περισσότερο από τη μισή από τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, περισσότερες μισές θα σταματήσουν. Ο χρόνος τελειώνει για το Ιράκ. Κατεπίγουσα ανάγκη μπορεί να σώσει το Ιράκ και το λαό της. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο σελίδα savepavlairak.info. μικρόφωνο, Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. σε κάποιες, από τους, κάποιους καταβλισμούς κοντά στο Ερμπίλ έχω πάει και στην Ιορδανία γνωρίζω και την κατάσταση στο Λίβανο στην Τουρκία και βλέπουμε ότι είναι εξαιρετικά απάνθρωπη η κατάσταση αυτή για τους ανθρώπους που είναι υποχρεωμένοι να ζουν εκεί. Αυτό δείχνει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Ότι ένα είναι η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά κάτι ξεχωριστό είναι η μόνιμη λύση. Γιατί τι κάνουμε στους καταβλισμούς, τα συμπτώματα αντιμετωπίζουμε, όχι την αιτία. Γι' αυτό ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να ακούσουμε τον κύριο Σαλίμ Αμπτούλα Αλκαβούρη, πρόεδρο της Βουλής του Ιράκ. Αλτζαμπούρη ως πρόεδρος της Βουλής και από την ε, πολιτική του διαδρομή έχει αποδείξει ότι εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή για να σταθεροποιήσει το Ιράκ που είναι προϋπόθεση για να επιτύχει η δική μας βοήθεια. Πρόεδρε Αλτζαμπούρη, έχετε το λόγο.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 بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس لجنة العلاقات في البرلمان ايش το όνομα του φιλέσλαχνου παντοδύναμου Θεού, κύριε ε, Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να λάβω το λόγο ενώπιό σας ε, εν ώψη του σχεδίου αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης στο Ιράκ. Θέλω να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος μου, εξ ονόματος του λαού μου καθώς και της κυβέρνησης του Ιράκ για ε, τη διοργάνωση αυτής της συνεδρίασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα των Ηνωμένων Εθνών υπό την προεδρία της κυρίας Λίσκα Καράντη που εργάστηκε πάρα πολύ ε, σκληρά Θέλω να ευχαριστήσω ε, όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που εργάζονται στο Ιράκ για τις τεράστιες προσπάθειες που μας βοηθούν να ανακουφίσουμε κάπως ε, τους εκτοπισμένους, ε, τους μετανάστες και τα θύματα της τρομοκρατίας. Ερχόμαστε από το Ιράκ που είναι το λίκνο του πολιτισμού. Σήμερα είναι σε ικτρή κατάσταση. Βλέπει μια τεράστια αιματοχυσία του λαού λόγω και εξαιτίας ε, αυτής της μεγάλης τρομοκρατικής επέλασης ε, που έχει πλήξει το λαό, του θεσμούς, το ίδιο το μέλλον της χώρας. Και ε, διακυβεύεται πραγματικά το μέλλον. Σήμερα το Ιράκ στέκεται όρθιο και πολιτικά και ο λαός με το κεφάλι ψηλά για να αντιμετωπίσει αυτή τη διεθνή τρομοκρατία που δεν απειλεί μόνο ε, το Ιράκ, ούτε πλήττει μόνο το Ιράκ αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Η τρομοκρατία ούτε σύνερο γνωρίζει, ούτε εξαιρέσει κάνει στο πρόγραμμά του. Ε, και αυτό θα πρέπει να είναι τεράστια η διεθνής προσπάθεια, οι διεθνείς οργανώσεις να συνεργαστούν μαζί μας και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να τερματιστεί αυτή η τρομοκρατία να μην τους επιτρέψουμε να ασκούν πιέσεις στους λαούς μας και να επιβάλλουν ε, ένα άλλο τρόπο ζωής στην κοινωνία μας. Η αντιμετώπιση, η πάταξη της τρομοκρατίας τελικά σημαίνει επένδυση στο μέλλον του λαού μας, των παιδιών μας, των κοριτσιών, των αγοριών για να ζουν με αξιοπρέπεια ε, βάσει και της διεθνούς συνεργασίας. Οι διεθνείς οργανώσεις εργάζονται κυρίως βάσει δωρεών, εξαρτώνται από δωρεές. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους δωρητές, όλους τους ενεχομένους για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι τώρα για να βοηθήσουν τους εκτοπισμένους και ιδιαίτερα άνδρες, γυναίκες, παιδιά, χείρες, χείρους, ηλικιωμένους, κάθε κατηγορία του πληθυσμού που ε, καταπιέζονται και καταπατώνται κατάφορα τα ε, δικαιώματά τους. Μπορεί κανείς να μιλήσει για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η αλληλεγγύη και η γενοδορία των δωρητών βοήθησαν λίγο να ανακουφιστεί ε, η ε, κατάσταση, ο πόνος και τα δεινά και σώθηκαν ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ανδρών, γυναικών, παιδιών, με φάρμακα, τρόφιμα, με παιδεία, σε αυτές τις τόσο περίπλοκες συνθήκες γίνεται μάθημα. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω μια έκκληση στην διεθνή κοινότητα να μην χαλαρώσει τις προσπάθειες για τη γενεοδορία και να απαντήσει θετικά ε, στην έκκληση αυτή. Έχει επιδεινωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις ε, ε, στο Ραμάντι, στην επαρχία της Αμβάρα. Σήμερα η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε υπερβαίνει τις δυνατότητές μας. Το Ιράκ καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ήταν κράτος δωρητής που υποδεχόταν όλους τους πρόσφυγες. Όποιον είχε ανάγκη το δεχόμαστε, τον υποδεχόμαστε ε, για βοήθεια, για παιδεία, για ε, ε, σύντηση. Σήμερα όμως βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Έχει μειωθεί και η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, οπότε η χώρα μας δεν δύναται να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εκατομμυρίων εκτοπισμένων. Ούτε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία του Ισλαμικού κράτους. Με τέτοια σφοδρή βία που υπερβαίνει κάθε φαντασία και κάθε ε, νόμο παραβιάζει, θεϊκό και ανθρώπινο του ματέου του του κόσμου. Εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν για να βοηθηθούν οι εκτοπισμένοι με ειδικές επιτροπές για να παρακολουθούν την κατάσταση των εκτοπιστέντων και όσων πλήττονται από τη βία για να έχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες. Το Ιράκ έχει εγκρίνει συνολικά σχέδια αποκατάστασης των περιοχών που απελευθερώνονται από την τρομοκρατία και τη μέγενη αυτή. Μπορούμε να βοηθήσουμε τις πόλεις να υποδεχθούν και πάλι τους κατοίκους τους. Έχουμε ένα κεντρικό κέντρο επιχειρήσεων 24 ώρες το 24ωρο. Ε, πυρετοδός εργάζεται για να παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές ε, σε κάθε Υπουργείο υπάρχει μονάδα ε, σε συναγερμό και ε, σε κάθε επαρχία με ε, πρόεδρο τον έπαρχο. Σε καθημερινή βάση λοιπόν παρακολουθούμε την κατάσταση και σε επίπεδο κυβέρνηση και σε επίπεδο κοινοβουλίου. Η κατάσταση κυρίες και κύριοι που αντιμετωπίζουμε σήμερα βαίνει επιδεινούμενη από μέρα σε μέρα και ε, τα δεινά που υφίστανται οι ε, κάτοικοι του Ιράκ είναι αντίστοιχα. Απευθύνω λοιπόν έκκληση προς τις δωρήτρες χώρες. Χρειαζόμαστε επιγόντως βοήθεια για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμά μας. Ο κίνδυνος της τρομοκρατίας δεν απειλεί μόνο τα άμεσα θύματα της, αλλά δεν γνωρίζει σύνορα. Κινδυνεύουν όλες οι κοινωνίες. Θα ήθελα να αποτίσω ένα φόρο τιμής και πάλι στις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, ιδιαίτερα τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Ιράκ. Έχουν εργαστεί σε συνθήκες ε, πραγματικά ιδιαίτερα επικίνδυνες όσο και και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τους εκτοπισμένους και μάλιστα σε πάρα πολύ απομακρυσμένα και ε, δυσπρόσιτα σημεία. Ευχαριστώ και πάλι όλες τις οργανώσεις και σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Thank you very much, President. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον Άντωνη Λέικ που είναι εκτελεστικός διευθυντής της ε, UNICEF. Ευχαριστώ πολύ όλους, τον κύριο Στυλιανίδη και όλους. Δεν ακούγεται στοιχώς ο μιλητής. Did anybody hear me? Καλώ uh, Καλώς, θέλω να ξεκινήσω και να πω κάτι που είναι κάπως ευχάριστο. Καλά, ναι. Το Ιράκ δεν έγινε όπως φοβόμαστε όλοι, μια λησμονημένη κρίση, ενώ ο κόσμος εστιαζόταν σε άλλες Ιράξεις κατά επίγουσες ανάγκες στον κόσμο. Πράγματι καθημερινά βλέπουμε το Ιράκ στους τίτλους των εφημερίδων, στις ειδήσεις τηλεοράσεις, στις συζητήσεις και στα κοινωνικά μέσα. Αλλά τα κακά μαντάτα είναι ότι οι τίτλοι, οι συζητήσεις, τα blogs πολύ συχνά συζητούν στατιωτικές και πολιτικές συγκρούσεις περισσότερο παρά την ανθρώπινη σφαγή και τα θύματα που έχουν δημιουργήσει. Σχεδόν ένα, πριν από ένα χρόνο είχε παγώσει ο κόσμος από βλέποντας ε, εκατοντάδες χιλιάδες να προσπαθούν να ξεφύγουν από τη Μοσούλη την, τα προβλήματα των Ιεζίντι και των άλλων μειονοτήτων και τα, οι γυναίκες και τα παιδιά που επολούντουσαν αγαθά στις αγορές Ακούγαμε ε, ιστορίες για σεξουαλική βία, για δολοφονίες. Σήμερα τέτοια προσοχή ε, λείπει ακόμα και αν αυξάνονται οι ανθρωπιστικές ανάγκες και συνεχίζονται οι φρικαλαιότητες. Και τώρα και τις επόμενες μέρες θα πρέπει να ακρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά το μέγεθος της κρίσης. Μια κρίση που δεν φαίνεται να έχει τέλος. Πρώτα απ' όλα ας δούμε κάποιους αριθμούς. Όπως είπε και ο κύριος Τηλιανίδης, πάνω από 8 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ιράκ και η μισή είναι παιδιά, χρειάζονται κατεπίγουσα βοήθεια. 8 εκατομμύρια. Φανταστείτε για μισό λεπτό έναν αριθμό ανθρώπων πέντε φορές το, το μέγεθος του πληθυσμού του κέντρου των Βρυξελών να χρειάζεται αυτά τα πράγματα είναι ανάγκη. Τον τελευταίο μήνα και μόνο πάνω από 200.000 άνθρωποι ε, έπρεπε να ξεφύγουν το Ραμάντι και αν, δεν, και αν δεν αρκούσε αυτό 250.000 πρόσφυγες από τη Συρία ε, προσπάθησαν να φιλοξενηθούν και να ξεφύγουν και να φιλοξενηθούν στο Ιράκ. Και η περιοχή του Κουρδιστάν φιλοξενεί περίπου ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπιστέντες ανθρώπους και πρόσφυγες. Αυτά δεν είναι στεγνά στατιστικά στοιχεία. Μιλάμε για ανθρώπους εδώ, μιλάμε για νούμερα. Ανθρώπους σαν αυτούς που είδαμε στην ταινία είναι οικογένειες που ξεριζώθηκαν τα σπίτια τους, από τις δουλειές τους, από τις ζωές τους, από τις κοινότητές τους. άντε και γυναίκες που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα καθημερινά και να προστατεύουν τα παιδιά τους και να τα κρατάνε ε, σε υγεία, να, να είναι χαρούμενα τα παιδιά τους. Παιδιά που θέλουν απλώς να παίξουν και να μάθουν. Αυτή η κρίση πρέπει να θυμηθούμε δεν πλήττει μόνο τους εσωτερικά εκτοπιστέντες και τους πρόσφυγες. Επίσης δοκιμάζει ε, και την δυνατότητα και τη γενοδορία των κοινοτήτων που φιλοξενούν αυτούς τους προσφυγές, των κυβερνήσεων, των ανθρωπιστικών οργανώσεων που φιλοξενούν, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν κλιμακούμενες ανθρωπιστικές ανάγκες και προσπαθούν να πλησιάσουν αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Διότι όλο και περισσότερο είναι δύσκολη η πρόσβαση. Πολλές από τις περιοχές τις οποίες εργαζόμεθα ελέγχονται από ένοπλες ομάδες. Και πέραν αυτού, ο ρυθμός και η μη προβλεψιμότητα των αναγκών η ανθρωπιστική κατάσταση αλλάζει, η ασφάλεια αλλάζει καθημερινά και πάρα πολλοί άνθρωποι μετακινούνται καθημερινά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους δώσουμε βοήθεια. Ακόμα χειρότερα βλέπουμε αρκετά ξεκάθαρα στον ορίζοντα εκατοντάδες χιλιάδες νέους εσωτερικά εκτοπιστέντες που πιθανότατα θα έρθουν διότι συνεχίζονται οι μάχες. Αλλά ακόμα αντιμετωπίζοντας αυτές τις περιστάσεις θα πρέπει να ενθαρρυνθούμε από τη διαφορά που κάνουμε εμείς και μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Συνεπώς, μαζί οι ανθρωπιστικοί εταίροι υποστήριξαν την κυβέρνηση για την παροχή τροφίμων, υδάτο και βασικών υπηρεσιών υγιεινής πάνω από 2 εκατομμύρια. Έχουμε 30 καταβλισμούς κατασκευαστήκαν από τον Ιούλιο πέρσι και στεγάζουν πάνω από 240.000 ανθρώπους και 13 άλλοι καταβλισμοί κατασκευάστηκαν για να καλυφθούν οι ανάγκες. Είχαν περιπτώσεις πολυμελίτιδας, έγιναν εμβολιασμοί σε 5,3 εκατομμύρια παιδιά και μια νέα εθνική εκστρατεία ολοκληρώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Ξεσημείω το αποτέλεσμα, αν δει κανείς τη μαζική μετακίνηση του πληθυσμού και την περίπλοκη κατάσταση να την ασφάλεια. Περίπου 270.000 εκτοπιστέντε παιδιά τα περισσότερο είναι τα πιο αθώα θύματα της σύγκρουσης και τα παιδιά είχαν κάποια πρόσβαση σε κάποιο είδους εκπαίδευση. Και αυτά τα κέρδη που ήταν πολύ δυσχεροί, αυτές οι επιτυχίες κινδυνεύουν, διότι υπάρχει τεράστια ανάγκη για ενίσχυση και βοήθεια και η δυνατότητα εμεί να ανταποκριθούμε είναι ανεπαρκή όσον αφορά τη χορήγηση τη βοήθεια. Είναι απλώ ανεπαρκή. Περίπου 4,4 εκατομμύρια άνθρωποι, επαναλαμβάνω, 4,4 εκατομμύρια χρειάζονται επισητιστική βοήθεια. Πάνω από 3 εκατομμύρια παιδιά σε και, και έφηβοι σε ηλικία παιδεία σχολείου δεν έχουν ε, την παιδεία. 650.000 και το παιδιά έχασαν σχεδόν ολόκληρη σχολική χρονιά. Πάνω από 7 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται νερό, χρειάζονται ε, υγειονομική περίθαλψη ε, και υπάρχουν και ασθένειες που, που, επιφυλα, που, επι, ε, που τους απειλούν η χολέρα, ε, η παροτίτιδα, είναι γενικά απειλές. Ας μην λησμονούμε τη φοβερή την απειλή από τη βία που αντιμετωπίζουν παιδιά και γυναίκες που αντιμετωπίζουν φυσική βιοπραγία, δουλεία, σεξουαλική βιοπραγία. Εγώ με φρίκι λέω ότι η σκλαβιά μεταξύ όλων αυτών, τη δουλεία, το λέω με φρίκι, όλα αυτά συνέβησαν και συμβαίνουν. Χρησιμοποιήθηκαν σαν ε, ε, ε, ε, ανθρώπινες ασπίδες και σαν άνθρωποι σαν, ε, για επιθέσεις αυτοκτονίας. Κάθε φρικαλαιότητα δεν επιτίθεται μόνο κατά των παιδιών που υπάρχουν, αλλά κατά το μέλλοντα. Ο συνδυασμό τη κακή διατροφή και ανεπαρκού υγιεινή περίθαλψη, η έλλειξη παιδεία και η βιοπραγία θέτει εν κινδύνο μια ολόκληρη γενιά νέων παιδιών. Διότι χωρί υγιή σώματα καινού, χωρί τα εργαλεία να ξαναφανταστούν ένα νέο μέλλον, χωρί την επιθυμία να συγχωρήσουν και να συμφιλειωθούν, πώ μπορούν να οικοδομήσουν το Ιράκ μετά το πέρα αυτή τη σύραξη με τόσε πολλέ προκλήσει και τόσε ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, θα ήταν πολύ εύκολο να αποκαρδιωθεί κανεί. Αλλά θυμάμαι τη διαφορά μεταξύ του να κάνει κανείς 70% των δεόντων και 80% των δεόντων. Αυτό αφορά τη ζωή και την ευημερία εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών και οικογενειών. Αλλά όπως θα μας πει η Λις Γκραντ, χωρίς συμπληρωματικού πόρους, πάνω από μισές από τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο Ιράκ θα σταματήσουν ή θα περικοπούν ε, τους επόμενους Αυτή Συνεπώς είναι μια κατεπίγουσα έκκληση. Πόσο επίγουσα τα τρόφιμα ήδη έχουν μειωθεί στην περιοχή του Νταχούκ, μια περιοχή που έχει το μεγαλύτερο αριθμό εσωτερικών εκτοπιστέντων, σε μισέ δόσει από εκείνου που ζουν εκτό των ε, καταβλισμών. Και οι περικοπέ θα συνεχιστούν αυτό το μήνα. Οι υπηρεσίε για νερό και υγεία στου εσωτερικά εκτοπιστέντε μειώνονται ε, και άλλε βασικέ υπηρεσίε. Αυτό έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, διότι πιο θερμοί μήνε προσεγγίζουν και εκεί έχουμε ε, το μεγαλύτερο κίνδυνο να ξεσπάσουν διάφορες ασθένειες με τη ζέστη. Παρά τις ε, ανάγκες αυτές πρέπει να είμαστε και πραγματιστές. Ξέρουμε ότι οι γενικές ανθρωπιστικές ανάγκες στον κόσμο αυξάνονται ενώ μειώνονται και είναι περιορισμένοι μάλλον ανθρώπινοι οι παγκόσμιοι πόροι. Γι' αυτό περικόψαμε αρχική μας έκκληση στα μισά και την περικόψαμε και την έκκλησή μας ξανά, αυτά που ζητούσαμε. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, είναι πιο κρίσιμη αυτή η έκκληση που απευθύνουμε. Χωρίς 500 εκατομμύρια δολάρια για το επόμενο εξάμενο, οι επιχειρήσει μα θα είναι στο, όριο του να καταρρεύσουν. Και δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτό να συμβεί. Δεν μπορούμε να μην ανταποκριθούμε στι ανάγκε του γενναίου λαού του Ιράκου που πολεμά κάθε μέρα για την επιβίωσή του. Κάθε μέρα που συναντούμε κάποιου από αυτού, κάθε φορά που βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των εσωτερικά εκτοπιστέντων, θυμόμαστε τι ψυχολογικέ προκλήσεις, οι φυσικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Όταν επισκέφτηκα την περιοχή Ανκάβα του Ερμπίλ στις αρχές του Ιανουαρίου, το είδα, ήταν, είχαμε ένα εμπορικό κέντρο που ήταν ημιτελές και βρήκα μια οικογένεια που προσπαθούσε να ξεφύγει και να βρει στέγη εκεί. Ήταν ο άντρα, η έγκυο γυναίκα, ένα, μια ηλικιωμένη τυφλή μητέρα και τρία παιδιά που έφτασαν ε, ένα μήνα πριν μετά που περπατήσαν τέσσερι μέρε για να φτάσουν εκεί. Παρά τι δύσκολε. Ε, ε, συνθήκε, ήταν πολύ περιορισμένο χώρο, δεν είχαν προστασία ιδιωτική ζωή και είχαν πολύ λίγο φα. Ήταν ευγνώμονε για την βοήθεια που έλαβαν. Διότι είχε γεννηθεί με ασφάλεια εκεί η δεύτερη κόρη του ζευγαριού και μου λέει ο σύζυγο, αυτό δεν είναι τίποτα να το συγκρίνει με αυτά που αφήσαμε πίσω μα. Το μόνο που χαιρόμαστε, είμαστε εδώ βλέπετε ασφαλείς. Το έχω ακούσει επανειλημμένα από το σχόλιο και υπογραμμίζει πόσο κρίσιμε είναι οι προσπάθειέ μα. Δίνουμε στου λαού του Ιράκ και τη Συρία όχι μόνο βοήθεια, του δίνουμε και ελπίδα. Παρόλα αυτά τα οποία πέρασαν, η οικογένεια, όπω τι άλλε οικογένειε, εξακολουθούν να έχουν ελπίδα. Για αυτού έχουν ελπίδα, για το Ιράκ έχουν ελπίδε, για την περιοχή και για το μέλλον μα. Διότι έχουμε ένα κοινό μέλλον. Γι' αυτό η βοήθεια που ζητάμε σήμερα δεν είναι για τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, η βοήθεια που ζητάμε είναι ώστε εμεί και τα Ηνωμένα Έθνη να βοηθήσουμε και τι οικογένειε και εκείνα τα παιδιά να κρατήσουν ζωντανέ τις ελπίδε του. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε την ε, δόκτωρα Μάγκαρα Ιτσάν που είναι ε, Γενική Διευθύντρια του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπρόκ, κύριε Μάκαβαν, κύριε Πρόεδρε της Ιρανικής Βουλής, κύριε Πίτροπε ε, Στυλιανίδη, ε, σας χαιρετώ και ευχαριστώ και ε, την αδελφή κυρία Χάν και τον αδελφό κύριο Λέικ. Ε, ε, Ακούσατε σήμερα το πρωί σειρά τρομακτικών στατιστικών στοιχείων που περιγράφουν ε, την απόγνωση ε, του Ιρακινού λαού. Και οι ε, προηγούμενοι προλαλήσαντες το περιέγραψαν πάρα πολύ εύγλωτα, το είδατε και στην ταινία. Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη και επιδεινώνεται ταχύτατα θρησκευτικές εντάσεις και ένοπλη σύραξη ε, κλείνουν πόρτες και ευκαιρίες για εκτοπισμένους πληθυσμούς να βρουν ε, ασφαλή ε, καταφύγια. Η πρόσβαση στην στοιχειώδη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι απόλυτη ανάγκη, αδύρυτη για 7 εκατομμύρια ανθρώπους. 77 είναι τα κέντρα υγείας και τα σχέδια και εξυπηρετούν περίπου 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι εγκαταστάσεις υγειονομικές ε, γνωρίζουν υπερπληθυσμό, δεν έχουμε φάρμακα, δεν έχουμε ιατροφαρμακευτικό υλικό, ακόμα και σε μεγάλα ε, νοσοκομεία αναφοράς. 14 νοσοκομεία και πάνω από 160 εγκαταστάσεις υγειονομικές έχουν καταστραφεί ε, στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο και σε ορισμένε περιπτώσεις 45% όλων των επαγγελματιών της υγείας έχουν ξεφύγει για να διασωθούν, για να σώσουν τη ζωή τους. Θα ήθελα να τονίσω ότι το Διεθνές Ανθρωπιστικό ε, Δίκαιο που ζητεί την προστασία των επαγγελματιών της υγείας, ε, των ε, νοσοκομείων, των ασθενοφόρων θα πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλα τα εμπλεκόμενα, τα μαχόμενα μέρη. Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, νερού, αποχέτευσης, καταραίων, είναι πολλά τα λοιμώδη σήματα για τους εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους. Ο καύσωνας έρχεται να επιδεινώσει το κίνδυνο ε, της ε, ανθρώπινης αυτής ένδια Έχουμε δει περιπτώσεις τώρα περιστατικά ηλαράς που ε, ε, αναφέρουν και 18 επαρχίες. Η χολέρα είναι ενδημική και εμφανίζεται και αυξάνεται και η λαϊσμανίαση. Δύο περιστατικά πολιομιελίτιδας επιβεβαιώθηκαν και τερματίστηκε ε, ένα καθεστώς 14 ετών ε, του Ιράκ που είχε κηρυχθεί ελεύθερο πολιομιελίτιδας. Βλέπετε πως καταραίει όλο το σύστημα υγείας. Ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση ούτε στα πιο βασικά μέσα ε, πρόληψης, δηλαδή τον εμβολιασμό. Όπως γνωρίζουμε από πρώτερη ε, ε, εμπειρία, ο ιός της πολυεμιλιαίτιδας, όπως και άλλοι, είναι πάρα πολύ έξυπνοι και εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρέχουν οι πόλεμοι. Ο κόσμος ε, με χρόνια νοσήματα ε, όπως καρδιακά, διαβήτη και καρκίνο χρειάζονται ε, τακτικά φάρμακα. Για τους περισσότερους καταλαβαίνετε ότι έχουν διακοπεί οι θεραπείες. Η εθνική αλυσίδα παροχής βασικών φαρμάκων έχει καταρρεύσει. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν αλλά το πρόβλημα ε, που τους εμποδίζει είναι η ε, έλλειψη ασφάλειας, η μη πρόσβαση σε δρόμους, η έλλειψη ε, καυσίμων και οι διακοπές ρεύματος που ε, διακόπτουν τη ψυχρή αλυσίδα. Παρ' όλα αυτά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και οι εταίρες μας κάναμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση. Με εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε βασικά φάρμακα και ε, υπηρεσίες, ακόμα και εκεί που σοβεί ο πόλεμος. Έχουν εμβολιαστεί παιδιά, τα είπε μόλις ο Τόνι. Αλλά κυρίες και κύριοι, χωρίς τη χρηματοδότηση, για να μπορέσουν οι εταίροι μας να συνεχίσουν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, 84% όλων των προγραμμάτων υγείας και των κέντρων υγείας θα κλείσουν πριν τα τέλη Ιουνίου. Είμαστε ήδη στον Ιούνιο. Σκεφτείτε λίγο μια στιγμή τι σημαίνει αυτό για το λαό του Ιράκ. Μια έγκυος γυναίκα που προσπαθεί να γεννήσει με ασφάλεια ένα παιδί με πνευμονία και διάρρεια. Αυτές είναι αρρώστιες που μπορούν να είναι θανατηφόρες εάν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως. Κάποιος με υπέρταση που χρειάζεται το φάρμακό του για την πίεση για να μην πάθει εγκεφαλικό ή να μην πάθει καρδιακή προσβολή. Συν όλοι οι τραυματίες που χρειάζονται αντιμετώπιση των τραυμάτων ή τουλάχιστον παυσίπονα για σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια της υγείας στην περιφέρεια και γενικότερα. Μπορούν να εκδηλωθούν κρούσματα ε, ή δεν γνωρίζουν ε, ε, σύνορα. Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας θα ήθελα και πάλι να τονίσω. Ο λαός του Ιράκ χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια για το να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να καλύψουμε τις ανάγκες υγείας είναι ανθρωπιστική προϋπόθεση ε, ε, όχι μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και αποκατάσταση της χώρας. Είναι απλές οι επεμβάσεις και δεν είναι τόσο ακριβές. Πολλά μπορούν να γίνουν ε, για να ανακουφιστούν η ένδυα και η απόγνωση κυρίως όλων αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων. Δώστε τους παρακαλώ ελπίδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Dr. Τσάν. Νομίζω ότι από όλου του ομιλητέ ε, έχουμε συνειδητοποιήσει από αυτά που μα είπαν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δράσουμε άμεσα και όλοι εδώ θα σκεφτούν πολύ σοβαρά τις επιλογές που κάνουν διότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα κλείσουν τόσα πολλά ιατρικά κέντρα. Είναι επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να δράσουμε για ανθρωπιστικούς λόγους αλλιώς ε, θα πολλαπλασιαστούν θα περιστατικά θα πρέπει να ζήσουμε αυτό το βάρος στη συνείδησή μας. Θα ήθελα τώρα να ε, προβάλλετε την επόμενη παρουσίαση και να έρθει παρακαλώ η κυρία Λίζε Γκραντ στο βήμα. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Λίζε Γκραντ, είναι ε, αναπληρωτήρια ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα αρμόδια για την αποστολή ουνάμι του ΟΗΕ. επίση είναι συντονίστρια, ε, συντονίστρια συγγνώμη, για την ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράκ. Κυρία Γκραντ, ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλο άνθρωπο για να μα μιλήσει σήμερα και να μα πει τι μπορούμε να, σε τι μπορούμε να ελπίζουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, να χαιρετήσω τους διακεκριμένους προσκεκλημένους στη σημερινή εκδήλωση. Θα ήθελα ε, να κάνω μια επισκόπηση της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, θα βασιστώ σε μια παρουσίαση PowerPoint που έχετε στις οθόνες σας. Το βασικό ε, μήνυμα είναι ότι η ανθρωπιστική κρίση ε, είναι από τις πιο περίπλοκες και πιο ευμετάβλητες στον κόσμο. Έχουν αναφερθεί και οι συνάδελφοι σε αυτό επίσης. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια ζωτικής σημασίας τετραπλασιάστηκε τα τελευταία 12 χρόνια. Αυτό σας λέω ότι είναι ραγδαίες η εξελίξη, εξελίσσεται ταχύτατα η κρίση. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, επηρεάζει η κρίση ε, όλες ε, και τις 18 ε, διοικητικές επαρχίες της χώρας ο συνολικό αριθμό αυτών που χρειάζονται βοήθεια. Βλέπετε πού εστιάζονται οι ανάγκες. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κόκκινος κύκλος, τόσο περισσότεροι υπάρχουν που χρειάζονται άμεση ανάγκε. Ε, μεγαλύτερο Anbar. Έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπων που χρειαζονται αμεση βοηθεια επαρχια ανμπαρ εχουμε πανω απο ενα εκατομμυριο ανθρωπων που χρηζουν προστασία. Ε, στην Ίνεβα 1,3, στο Κίρκουκ 1,18 ε, και ούτω καθεξής. 8,2 εκατομμύρια ε, άνθρωποι συνολικά χρειάζονται ε, βοήθεια. Ξέρουμε ότι θα επιδεινωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση και το Μέχρι το τέλος του 2015 προβλέπεται ε, και άλλα 2 εκατομμύρια να ζητήσουν βοήθεια, δηλαδή συνολικά 10 εκατομμύρια ε, Ιρακινών, ε, ενώ ο συνολικός πληθυσμός είναι 36 ε, εκατομμύρια. Αυτά μας λέει το εφεδρικό μας σχέδιο. Επίσης, είναι εξαιρετικά περίπλοκη και ευμετάβλητη, πολυσύνθετη αυτή η κρίση του Ιράκ ε, και οι δυνατότητες ε, για το δυναμικό των ανθρωπιστικών οργανώσεων δοκιμάζεται στο Ιράκ. Είδατε τα τρομακτικά ταρατιστικά στοιχεία του Άντωνι Λέικ. Πάνω από 4,4 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται άμεσα τροφή. Επίσης, σε βασικές γεωργικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και τις μεγάλες ζώνες του Ιράκ που συνορεύει με τη Συρία ε, έχει σοβαρό επιστημιστικό πρόβλημα. Επίσης, ε, σε ολόκληρο το Ιράκ ε, ε, στεγάζονται σε, όπου μπορούν οι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Αυτό μας εμπνέει ιδιαίτερα, όμως ε, είναι μεγάλο το κόστος της γενεοδορίας του πληθυσμού. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες κοινότητες υποδοχής που ζουν αποθλειωμένοι διότι έχουν πέσει στην παγίδα της φτώχειας πάρα πολύ στο Ιράκ διότι έχουν υποδεχτεί στα σπίτια τους εσωτερικά εκτοπιστέντες το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Άντιν Λέικ και άλλοι που παρενέβησαν ε, μα είπαν ότι βρίσκεται στο χείλο του γκρεμού ε, η χώρα. Ε, πρέπει να το τονίσουμε αυτό επανειλημμένα θεωρούμε ότι αν καταρρεύσει η ανθρωπιστική αποστολή και αν δεν προκύψει νέα χρηματοδότηση αυτό θα συμβεί, η εθνική συμφιλίωση στο Ιράκ θα υπονομευθεί και περαιτέρω κερματισμός προβλέπεται. Είναι μεγάλα τα διακυβάγματα στο Ιράκ και τώρα χρειαζόμαστε αλληλεγγύη, αλληλεγγύη προς πολίτες και αλληλεγγύη προς την κυβέρνηση του Ιράκ. Πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό ε, στις ε, πρώτες παρεμβάσεις ότι οι από τις κατάφορες παραβιάσεις ε, των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημειώνονται στο Ιράκ ε, και είναι μια κρίση που χρειάζεται προστασία προς τον πληθυσμό που βρίσκεται εν κινδύνο. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό της κρίσης. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ολόκληρες γενιές νέων που κινδυνεύουν καθημερινά. Είπαμε επίσης ότι οι διαθρησκευτικές εντάσεις κλιμακώνονται και θέτουν εν κινδυνό την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 ε, θελοντική επιστροφή στις αιστείες τους των τριών εκατομμυρίων εστερικά εκτοπιστέντων. Βλέπετε ε, με σκούρο και μέσο μπλε ε, τις περιοχές όπου υπάρχει πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση και ακριβώς αυτές τις περιοχές θεωρούμε ότι μερικοί από τους πλέον ευάλωτους διαβιούν αυτή τη στιγμή. Αυτοί που θα έπρεπε να μας ανησυχούν περισσότερο είναι ακριβώς τις περιοχές που δυσκολευόμαστε πάνω απ' όλα να φτάσουμε. Και όποιος παρακολουθεί τις ειδήσει για το Ιράκ ξέρει ότι από ανθρωπιστική σε πλευρά τα πράγματα σίγουρα θα χειροτερεύσουν. Ε, είναι ε, το ε, καλοκαίρι της απόγνωσης, έτσι το ε, ονομάζουμε, τους επόμενους μήνες λόγω της ε, σύραξης ε, της, των εξεγέρσεων και αντεξεγέρσεων θα κλιμακωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες κατά 1,7 έως 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτές είναι οι προβλέψεις. Το εφεδρικό μας σχέδιο που τώρα συγκροτούμε μας λέει ότι μπορεί πολλαπλές κοινότητες και πολλαπλές πόλεις ταυτόχρονα να πληγούν από την κρίση και σε αστικές περιοχές, ε, ολόκληρες συνοικίες, όπως είδαμε στο Ραμάντι ε, την περασμένη εβδομάδα, ε, θα έχουν ως αποτέλεσμα να φεύγουν μαζικά οι άνθρωποι από τα σπίτια τους. Χιλιάδες, 70.000 άνθρωποι μέσα σε 48 ώρες έφυγαν από το Ραμάντι και τις προσεχείς εβδομάδες παρεμφερεί φαινόμενα θα παρατηρηθούν, όπως ακριβώς το Ραμάντι οι εταίροι μας για την ανθρωπιστική δράση καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και χάρη σε αυτούς ε, ε, θα ήθελα να χαιρετήσω αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μη κυβερνητικής οργάνωση, Ανθρωπιστική Οργανώσει, που είναι στην πρώτη γραμμή και παρέχουν τις υπηρεσίες τους όπως είπε ο Άντων Λέ και η Δόκτωρ ε, Τσάνε, πάνω από 150 οργανώσεις ε, έχουν ε, βοηθήσει περίπου το μήνα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους ε, το τελευταίο χρόνο και μιλώντας για τις επιχειρήσεις πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για τις προκλήσεις στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθουμε διότι κλιμακώνεται ραγδαία η κρίση και όπως σας είπα αγωνιζόμαστε, διότι είναι πολύ σύνθετη η κρίση, αγωνιζόμαστε γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες ε, και γι' αυτό τώρα ε, ε, μεταρρυθμίζουμε το, την, την επιχειρησιακή μας δομή και αναδιαρθρώνουμε το επιχειρησιακό μας κέντρο. Προσπαθούμε να φτιάξουμε νέους εδιάβλου, να του τροφοδοτούμε και να του έχουμε τοποθετήσει πρωτού προκύψει η κρίση. Διευρύνουμε τις εγκαταστάσεις αποθήκευση. Σα είπα ότι για ολόκληρη τη χώρα έχουμε ένα εφεδρικό σχέδιο που αναπτύσσουμε τώρα και φροντίζουμε να έχουμε όσο το δυνατόν γίνεται ακριβέστερα στοιχεία. Επίσης υπάρχουν συντονιστικοί μηχανισμοί ε, με την κυβέρνηση, του οποίου ενισχύουμε. Ένα από τα βασικότερα ζητήματα το έφυξε ήδη ο Άντωνι Λέικ όταν μας μίλησε για την ε, το μηχανισμό έγκαιρης ανταπόκρισης. Ε, δηλαδή μέσα σε 48 ώρες ε, ο ΙΕ με τους εταίρους με τις μη οργανώσεις προσφέρει στις οικογένειες ένα κίτ βοήθειας έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή τροφή για τις πρώτες μέρες, οτιδήποτε χρειάζονται μέσα σε ένα κουτί. Την επίγουσα ανάγκη και ο ΙΕ και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μετά φέρνουν μεγαλύτερα κουτιά για να μπορέσουν να στήσουν ένα ένα πρόχειρο σπιτικό και πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι σε 2.000 διαφορετικές ε, τοποθεσίες έχουν λάβει αυτό το κουτί πρώτης ε, βοήθειας. Ε, ποια είναι η μεγαλύτερη μας ανησυχία, ότι τελειώνουν αυτά τα κουτιά άμεσης βοήθειας τελευταίες εβδομάδες. Αν πέσει στην κατοχή του ίσης η αντίθεη Σαμάρα, μια άλλη πόλη, αν συμβεί κάτι τρομακτικό, θα βρεθούμε με αυτή την κατάσταση. Δεν θα έχουμε αυτές τις, αυτά τα κουτιά πρώτης βοήθειας, ζωτικής βοήθειας πέρα από το μηχανισμό έγκαιρης ανταπόκρισης είναι σημαντικό διότι σε ακραίες περιστάσεις μπορούμε να φτάσουμε, να φτάσει βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Μιλήσαμε για ζωφερή πραγματικότητα πάνω από 50% όλων των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων θα κλείσουν ή θα περικοπούν εάν δεν λάβουμε άμεσα χρηματοδότηση. Είναι ένα γεγονός αυτό. Δεν υπερβάλλω όταν το λέω, πρόκειται για συγκεκριμένα στοιχεία. 50% το ίμιση των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων θα κλείσουν ή θα περιοριστούν αν δεν λάβουμε χρηματοδότηση. Όπως είπε ο Άντωνη Λέιθε, το παγκόσμιο πρόγραμμα, ε, το επιστημιστικό έχει μειώσει ήδη ε, τις ε, ποσότητες ε, των δελτίων ε, και 77% των κέντρων κινδυνεύουν να κλείσουν όταν κλείνει ένα ιατρικό κέντρο, μία κλινική καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους θα κλείσουν άμεσα 77 ιατρικά κέντρα και σας είπα ότι τελειώνει το στόκ που έχουμε το απόθεμα από τα κουτιά ε, ζωτικής ε, ε, βοήθειας, άμεσης ανάγκης, για να ανακεφαλαιώσω τα βασικά ζητήματα. Η κυβέρνηση του Ιράκ ηγείται της επιχείρησης και έχει αναλάβει πλήρη δέσμευση και δραστηριοποιείται για τη διεξαγωγή της επιχείρησης. Κάνει μεταφορές μετρητών, δίνει στίγη, έχουν φτιάξει καταβλισμούς, έχουν ανοίξει τα ιατρικά κέντρα, τις ε, κλινικές και τα σχολεία. Όμως 40% του προϋπολογισμού χάθηκε ε, λόγω της μείωσης της τιμής ε, του πετρελαίου το περασμένο χρόνο και επίσης έχουν και την αντεπίθεση από τον Ίσιλ, είναι με την πλάτη στον τοίχο, δεν έχουν πόρους πλέον. Σε μια χώρα όπως το Ιράκ περιμένουμε να φέρει το βάρος της ανθρωπιστικής δράσης και όντως έκανε αυτό που της αναλογούσε η κυβέρνηση. Τώρα σας ξαναλέω τους έχουν στριμώξει στον τοίχο. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Χρειάζονται βοήθεια τώρα. Και γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση σε διεθνές επίπεδο και λέμε στην διεθνή κοινότητα τώρα πρέπει να καταδείξετε την αλληλεγγύη σας προς την κυβέρνηση και το λαό του Ιράκ. Ε, αυτό είναι το σχέδιο ε, ανθρωπιστικής έκτακτης βοήθειας. Ε, είναι η θερμότερη έκκληση που έχουμε απευθύνει στην περιοχή. Ξέρετε, όσοι ξέρουν τον ΟΗΕ περιμένουν κάτι με ψαχνό. το κάνουμε αυτό διότι προσπαθούμε να, έχουμε, να σεβόμαστε διεθνή ελάχιστα πρότυπα όταν παρέχουμε βοήθεια. Όμως όπως είπαν και οι συνάδελφοι ξέρουμε ότι ανά τον κόσμο. Υπάρχουν κρίσεις που πιέζουν ασφικτικά τους προϋπολογισμούς των δωρητών. Το ξέρουμε αυτό, δεν είμαστε αφελείς. Γι' αυτό σας είπαμε ότι στο Ιράκ σε κάθε ομάδα, σε κάθε κλάστερ θα δώνουμε ένα ελάχιστο πακέτο το οποίο ε, θα ταξινομείται ε, σε ε, ανταπόκριση πρώτης γραμμής, δεύτερης γραμμής και πλήρης κάλυψης. Πλήρους κάλυψης. Εμείς θέλουμε να απευθύνουμε μια, μια έκκληση που θα περνάει το εξή μήνυμα ότι κάνουμε κάθε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τηρήσουμε τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα. Δεν είμαστε όμως σε θέση να το κάνουμε αυτό. Οπότε ε, είναι αποστεωμένο το πρόγραμμά μας, αν θέλετε, διότι είναι το ελάχιστο πακέτο βοήθειας ε, που ε, υπακούει σε αυτές τις τρεις κατηγορίες σε ανταπόκριση πρώτης, δεύτερης γραμμής και κλάστερ, δηλαδή καλύπτοντας ολόκληρη όλες τις ανάγκες. Ως ε, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα διεθνή πρότυπα, διότι αυτή είναι η δουλειά όποιον αναλαμβάνει ανθρωπιστική δράση. Έχουμε περιορισμένο προπολογισμό, περιορισμένη πρόσβαση, περιορισμένο δυναμικό και είμαστε υποχρεωμένοι εκ των περιστάσεων να δώσουμε ένα ελάχιστο πακέτο βοήθεια και γι' αυτό ζητάμε τη βοήθειά σα 500 ε, εκατομμύρια δολάρια για τους επόμενους 6 μήνες, 2,6 ε, εκατομμύρια τους επόμενους μήνες, 2,6 ε, εκατομμύρια ανθρώπων συγγνώμη, 5,6 εκατομμύρια. Έχουμε ε, ως προς την διεθνή δέσμευση ε, ναι, μια ανάγκη εξισορρόπησης ε, για την ίδια κατανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχουμε πέντε στρατηγικούς στόχους, ειδικευμένη βοήθεια για την προστασία, διότι πρόκειται για επιχείρηση προστασίας, διατήρηση της βοήθειας σε ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, για αυτούς που μας χρειάζονται απολύτως και προσπαθούμε, ακόμη και αν δεν είναι σε κρατικά ελεγχόμενες περιοχές, να έχουμε πρόσβαση σε αυτούς τους ανθρώπους, βοήθεια βοηθώντας εσωτερικά ε, εκτοπιστέντες σε ολόκληρο το Ιράκ και το τελευταίο σημείο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια κοινωνική πλατφόρμα που θα βασίζεται σε μετρητά, ε, σε βοήθεια μετρητών, ε, σε συνεργασία με την ε, κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική εξόδου από την κρίση. Υπάρχει ένα γενναιόδωρο, μια γενναιόδωρη κοινωνική πλατφόρμα στο Ιράκ ήδη όμως αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένη στον τοίχο η κυβέρνηση και δεν έχει το επιθυμητό εύρος αυτή η πλατφόρμα, όμως θα ξανανεύει η τιμή του πετρελαίου και όταν συμβεί αυτό ε, δεν θα χρειάζεται οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να κάνουν αυτό που κάνουμε τώρα. Όμως προς το παρόν δεν ισχύει αυτό, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Θέλουμε όμως δηλαδή, να υποστηρίξουμε τη μετάβαση προς ε, μια κοινωνική πλατφόρμα που θα βασίζεται σε ματριτά. Αυτή είναι η στρατηγική εξόδου μας. Σας είπα ότι έχουμε το ελάχιστο πακέτο πρώτης, δεύτερης γραμμής και πλήρους ανταπόκρισης σε αυτήν τη σταδιακή προσέγγιση για να δώσουμε αποχέτευση πόσιμο νερό, τρόφιμα, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες, εμφιαλωμένο νερό, λοιπόν, τουαλέτες, σε σαπούνι και σε δεύτερο επίπεδο έχουμε αγγλίες, ε, υδροφόρες και ούτε καθεξής. Ε, υπάρχει παρακολούθηση και ε, προσπαθούμε να διευρύνουμε τα δίκτυα υδροδότησης και αποχέτευσης. Είναι 13 οι ομάδες, 13 τα κλάστερς και δραστηριοποιούμαστε εξίσου σε όλα και βλέπουν όλοι αυτή την προσέγγιση σε τρία βήματα που σας έλεγα. Τέλος... Ε, είναι η μόνη κρίση στον κόσμο επίπεδου 3 ε, που έχει μια ρεαλιστική στρατηγική εξόδου. Αυτή η κοινωνική πλατφόρμα που σας έλεγα που βασίζεται σε βοήθεια σε μετρητά. Ήδη σε συνεργασία με την κυβέρνηση προσπαθούμε να συμβάλλουμε και εμείς τόσο ώστε να αναβαθμιστεί αυτή η πλατφόρμα, ώστε να ε, μα λυθούν τα χέρια, μην χρειάζεται να κάνουμε εμείς αυτά που κάνουμε τώρα. Ποια είναι η έκκλησή μας λοιπόν, ε, ε, ε, αυτή είναι, σας είπα, η ευρύτερη και η πιο αποστεωμένη έκκληση σε διεθνές επίπεδο που υπήρξε ποτέ. προστασία 54 εκατομμύρια, επιστημιστική ασφάλεια 180, υγεία 60 εκατομμύρια, νερό, αποχέτευση και υγιεινή 43,9, σχεδόν 100 εκατομμύρια για τη στέγη και, την, και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες πέρα από την τροφή, 2,5 για τους καταβλισμούς, 26 για την εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Τα βλέπετε στους οθόνες σας θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας προς ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς ε, την Επιτροπή, την ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΟ, προς τον Επίτροπο και προς όλους όσους συνεργάστηκαν για τη σημερινή εκδήλωση. Επίσης, να ευχαριστούμε την κυβέρνηση του Ιράκ και την προσωρινή κυβέρνηση του Κουρδιστάν που μας δέχτηκαν στη χώρα και μας επιτρέπουν να δραστηριοποιούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σαφώς αναφερθήκατε στις ανάγκες, το κόστος αυτών και ελπίζω να καλύψουμε τις ανάγκες. Το επόμενο μέλος του πάνελ παρακαλώ να έρθει εδώ και θα αλλάξουμε θέσεις. Να έρθουν επόμενοι, τα επόμενα μέλη του πάνελ. Πρέπει να αποχωρήσω. Πρέπει να πάω στην Ευρωπαϊκή Μερίδα Ανάπτυξης που λαμβάνει η χώρα στις Βρυξέλλες όπως και άλλοι συνάδελφοι. Θα δώσω την Προεδρία. Σε συνάδελφο έχουμε υπόψη τα θέματα και θα τα συζητήσουμε και στην ημερίδα ανάπτυξη. Στον κύριο Περμόη θα δώσω το λόγο, αντιπρόεδρο της Επιτροπής ε, ΑΦΕΤ. Καλημέρα σας. Πάμε λοιπόν στο σημείο 6, που είναι το ανθρωπιστικό πια πάνελ. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Σόρενσεν, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΕΧΟ, για να μας ε, κάνει την εισαγωγή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Σόρενσεν. Ε, ε, Καλημέρα σε όλους. Γνωριζόμαστε. Ε, λοιπόν, λοιπόν, είμαι ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, ε, Κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, γνωριζόμαστε πολύ καλά. Από πλευρά ΕΚΟ, που είναι η Υπηρεσία ανθρωπιστική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά απόψή μα είναι μεγάλη ευκαιρία εδώ να τονίσουμε τι μαζικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουμε και τις διεξόδους που διαφαίνονται. Πρέπει να στεστούμε εις κατεπίγωσες ανάγκες για την προστασία των αμάχων. Πολλοί είπαν ότι είναι κρίση προστασίας αυτή και θέλουμε να δώσουμε και ανθρωπιστική βοήθεια βασική. Είναι πρόκληση όταν αντιμετωπίζουμε ανθρωπογενείς καταστροφές όπως αυτή. Και έχουμε και πολιτικά διακυβεύματα. Ολόθερμα υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Λίζα Γκραντ Όλοι εντυπωσιαστήκαμε από την παρουσίαση που έκανε. Ήτανε και ποιοτική. Και έμφερμη παρουσίαση. Και χάρη σε εκείνη και την υποστήριξη των διαφόρων φορέων και των εταίρων που είναι παρόντες στο Ιράκ, έχουμε θετική εξέλιξη όσον αφορά την ανθρωπιστική ανταπόκριση. Θέλουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ελεγχόμενη ανθρωπιστική δράση. Τι θα θέλαμε να τονίσουμε. Τρία βασικά χαρακτηριστικά της ανταπόκρισής μας. Θέλουμε γενική προσέγγιση ολιστική για το Ιράκ. Είναι εύκολο να εισαζόμαστε στις εύκολα προσβάσιμες περιοχές. Όμως ανέφεραν πολλοί ομιλητές ότι πολλοί λαοί, πολλοί κόσμος με ανάγκες βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν δέχτηκαν ανθρωπιστική βοήθεια τους τελευταίους μήνες. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Υπέχουμε ηθική υποχρέωση, όπως είπε και ο Επίτροπος, και ανθρωπιστική υποχρέωση, να πλησιάσουμε όλους τους έχοντες ανάγκες οπουδήποτε. Δεύτερο χαρακτηριστικό της απαντήσεως και της ανταποκρισίσεως που προτείνεται είναι ολοκληρωμένη προσέγγιση. κατεπηγόντως. Χρειάζεται ένα κέντρο ανθρωπιστικής βοηθείας στη Βαγδάτη και στο Ερμπίλ. Είναι ακρογωνιός λίθος για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες. Να υπάρχει σωστός συντονισμός του σχεδιασμού. Να διευκολυνθεί η διαπραγμάτευση για πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Χρειάζεται συντονισμός λοιπόν. Γίνεται σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης συντονισμός και σε άλλα επίπεδα. Θα ακούσουμε και τον Υπουργό για την ανθρωπιστική βοήθεια αργότερα. Και χαιρετίζουμε και το μηχανισμό ταχείας ανταπόκρισης είναι βασικό εργαλείο για ταχύ ολοκληρωμένη βοήθεια για τους έχοντες ανάγκες, τους εκτοπιστέντες σε δυσπρόσιτες περιοχές. Να καλυφθούν δραματικά κενά στην ανθρωπιστική βοήθεια. Τι εννοώ, να προληφθούν ε, απώλειες ζώων. Και τέλος, όπως αναφέρθηκε από τη Λίζ, Χρειαζόμαστε και πολιτική εξόδου, σωστή αυτή παρουσιάστηκε, αλλά χρειάζεται και συντονισμένη και εναρμονισμένη βοήθεια σε μετρητά και σχετικός μηχανισμός, οικονομική βοήθεια. Είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής. Εργαλείο που χρειάζεται για την ενοποίηση και ανοικοδόμηση του κοινωνικού ιστού στο Ιράκ που χρειάζεται για το μέλλον, για τη σταθερότητα της χώρας. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βασικές ανάγκες των πληγέντων πληθυσμών. Χρειάζεται πιο αξιοπρεπής αντιμετώπιση πέρα από τη διανομή τροφίμων και φαρμάκων. Δεν θα είναι εύκολο να εφαρμοστούν όλα αυτά. Χρειάζεται καινοτομία στην προσέγγιση ανθρωπιστική βοήθεια. Χρειάζεται προσπάθειες όχι πλευρά δωρητών μόνο, αλλά και από τις επιτόπιου φορείς και από τις δημόσιες αρχές στο Ιράκ. Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τις προσπάθειες και σαν δωρητέ θα συμμετάσχουμε στην εφαρμογή του προγράμματος αυτού παροχής οικονομικής βοήθειας. Με τα χαράς θα επανέλθω στη συζήτηση που ακολουθήσει. Ευχαριστώ κύριε Σόρενσεν. Έχουμε υψηλού επίπεδου ε, πάνελ. Ε, είναι πάρα πολύ εξέχουσε ε, προσωπικότητε και θα του δώσω μέσα το λόγο. Είναι πρώτο ο κύριο Φόλκερ Τούρκ που είναι ο ύπατο εκπρόσωπο, ε, αναπληρωτή μάλλον ύπατο εκπρόσωπο ε, για του πρόσφυγε, τη ύπατη αρμοστία. Ευχαριστώ ε, πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση. Όπως είπαν οι προλαλήσαντες κυρίως η Λίς Γκράντε, είναι μια κρίση πραγματικά προστασίας και χαίρομαι που ε, έχω την ευκαιρία ως αρμόδιος για την προστασία να σας πω κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αν κοιτάξουμε τις στατιστικές, ε, είδαμε πολλές στατιστικές ε, μιλάμε για εκατομμύρια, πάνω από 8 είναι αυτοί που έχουν ανάγκη. Ε, υπάρχουν πολλοί μετατοπισμένοι, εκτοπισμένοι, 3 εκατομμύρια σχεδόν ε, τη τελευταία διετία. 900.000 προηγουμένως είχαν εκτοπιστεί και ήρθαν να προσθεθούν σε αυτούς και ο συνολικός πληθυσμός αγγίζει τα 4 εκατομμύρια αν προσθέσετε και 185.000 πρόσφυγες από το Ιράκ που έχουν μεταβεί σε γειτονικέ ε, χώρες ή ακόμα πιο μακριά. Ε, είναι πολύ ε, σημαντικό αυτό, πολύ ισχυρό και όπως γνωρίζουμε τι σημαίνει ο εκτοπισμός, φτωχοποίηση της κοινωνίας και των ίδιων των ανθρώπων που πλήττονται άμεσα. Αν κοιτάξουμε τον κάθε άνθρωπο ε, που είναι πίσω από τους αριθμούς, άντρα, γυναίκα, παιδί, είναι τραγωδίες και πολλές φορές είναι πολλαπλός ο εκτοπισμός γιατί είναι ακόμα ένα φαινόμενο στο Ιράκ. Οι άνθρωποι αυτοί εκτοπίζονται επανειλημμένα. Δεν ε, είναι στις αιστείες τους αυτοί που εκτοπίζονται. Ήδη στο παρελθόν έχουν εκτοπιστεί, έχουν φτωχύνει και τώρα ξανά εκδιώκονται. Είμαστε σε πάρα πολύ τραγική κατάσταση. Αν δείτε τις καταγραφές ε, και τις απογραφές είναι πραγματικές τραγωδίες και τραυματικές καταστάσεις με άκρα βία και σεξουαλική βία κακοποίηση σε πολύ κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ε, αν βρούνε κάπου ένα ασφαλές καταφύγιο, αν βρουν, γιατί είναι και σε πολιορκία πολλές φορές ο πληθυσμός, σε περίπτωση που βρεις ένα ασφαλέ καταφύγιο, είναι πάρα πολύ σχετική αυτή η έννοια της ασφάλειας. Όποιος ασχολείται με την διάσταση της προστασίας, ε, καταλαβαίνει ότι η ανθρωπιστική απάντηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρή, πάρα πολύ γερή ε, και να απαντά στις ανάγκες των ανθρώπων αυτών των ίδιων και τα όσα εκείνοι ζητούν. Θα ήθελα να πω συγκεκριμένα το εξή. Ε, μόλις είχα την ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή Ελευθεριών τη ΛΥΜΠΕ ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μπορεί να νομίζετε ότι δεν υπάρχει μεγάλη σύνδεση. Υπάρχει όμως. Τι μάθαμε από το παράδειγμα της Συρίας. Ότι πολλοί Σύριοι τώρα φτάνουν στα πλοιάρια και προσπαθούν να ε, διασχίσουν τη Μεσόγειο, ιδιαίτερα από την Τουρκία στην Ελλάδα. Αυτό δεν το είχαμε δει για κάποιο διάστημα. Ε, ακριβώς επειδή ε, διαιωνίζεται η σύραξη, ε, αναγκάζονται και οι Σύροι να φτάνουν στη Μεσόγειο και στις χώρες που εσείς εκπροσωπείτε. Θα δούμε λοιπόν αντίστοιχο φαινόμενο και με Ιρακινούς. Ήδη έχουμε δει Ιρακινούς που προσπαθούν να περάσουν από τη Τουρκία στην Ελλάδα. Οπότε θα πρέπει η απάντησή μας, η απόκρισή μας να είναι ξεκάθαρη. Τι ανάγκες υπάρχουν ανθρωπιστικές εντός του Ιράκ, αλλιώς ο κόσμος θα φύγει αν δεν δεχτεί την υποστήριξη που χρειάζεται. Θα προσπαθήσει να βρει αλλού τη μοίρα του. Ε, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στο Ιράκ οι ίδιοι. Είναι σημαντικό δίδεγμα αυτό και από τη Συρία αλλά και ε, αν το συνδέσουμε με το, τα όσα βλέπουμε να εκτελήσουν μπροστά στα μάτια μας στη Μεσόγειο. Κάτι που επίσης είπε η Λις Γκράντε και έχει σημασία, το είδα και εγώ η διεισόμαση όταν είχα πάει σε αποστολή στο Ιράκ πριν από λίγες εβδομάδες, υπάρχει ένα τεράστιο αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης, όπως είπε και ο Τόνι Λέικ, δείχνουν τη μία εικόνα, αυτή τη ζωφερή, τη στρατιωτικοποίηση, την ένοπλη σύραξη, τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει και άλλη ιστορία να διηγηθεί κανείς ε, η διαπροσωπική αλληλεγγύη των ίδιων των Ιρακινών μεταξύ τους. Αυτό είναι τεράστια σημασία συστατικό για όποια μοίρα επιφυλάσσει το μέλλον στο Ιράκ. Θα πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή την αλληλεγγύη άνθρωπος προς άνθρωπο με πάρα πολύ συγκεκριμένη προστασία. Για παράδειγμα είχα την ευκαιρία εγώ να συναντηθώ με κάποιους έξω από το Ερμπίλ που είχαν φτιάξει μια κοινότητα και υποδέχοντα ακόμα και Σύρους πρόσφυγες που είναι 250.000 περίπου, 250.000 ιδιαίτερα στις κουρδικές περιοχές εκεί γύρω από το Ερμπίλ ε, συγκεντρώθηκαν, έφτιαξαν μια κοινότητα προσπαθώντας να ε, λύσουν μόνοι τους κάποια από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Ακόμα και τα θέματα ε, της εκπαίδευσης των παιδιών, των ε, εξαναγκαστικών γάμων, της απογραφής τους κτλ. Δηλαδή, μπορούμε να βασιστούμε σε δομές υφιστάμενες, κοινωνικές, ένα δίκτυο υποδομών που υπάρχει των κοινοτήτων μεταξύ των ανθρώπινων. Εκεί θα πρέπει να οικοδομήσουμε και το μέλλον του Ιράκ. Είναι επένδυση ε, στο ανθρώπινο δυναμικό. Ήδη προετοιμάζεται το μέλλον και υπάρχει ο σπόρος για ένα πιο ειρηνικό μέλλον στο Ιράκ. Από τη δική μας σκοπιά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε την ευκαιρία στις κοινότητες αυτές να βοηθηθούν οι ίδιες με την ανθρωπιστική χρηματοδότηση που τόσο επιγόντως έχουν ανάγκη υπάρχει μια στρατηγική εξόδου ε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γίνεται γιατί δεν μπορούν οι αρχές της χώρας να αναλάβουν ε, τις τύχες τους. Δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και είναι ε, προς όφελος του άμαχου πληθυσμού αυτού, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο θύμα. Και ένα τελευταίο, να προτείνω κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα λύσεις για τους εκτοπισμένους. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα και θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα. Ε, και θα αυξηθεί ο εκτοπισμός μετά από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ακούμε ότι θα υπάρξουν ε, εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένων ε, στους επόμενους μήνες ε, πριν τα τέλη του έτους αλλά θα δούμε και επαναπατρισμούς, επιστροφές στις αιστείες σε κάποιες κοινότητες ορισμένων ή επανεγκατάσταση στο εσωτερικό του Ιράκ, δηλαδή θα εντάσσονται σε υφιστάμενες δομές και κοινότητες. Εμείς θα πρέπει να το υποστηρίξουμε με βάση τις αρχές που απαιτεί η προστασία. Δηλαδή θα πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση, να παρακολουθήσουμε, να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη, δυναμική του πληθυσμού και των μετακινήσεων. Και χρειάζεται πραγματικά ενεργή, ε, ενεργός υποστήριξη για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στις αιστείες τους με κάποια αξιοπρέπεια ή όταν μετεγκαθίστανται να έχουμε υπόψη μας τη συνολικότερη εικόνα. Οπότε μπορούμε να πούμε με τα λόγου γνώσεως ότι αυτά που βλέπουμε να τεκταίνονται στο Ιράκ σήμερα και στην ευρύτερη περιοχή είναι αλληλένδετα και με τα όσα διαδραματίζονται στην Ευρώπη. Και με τη χρηματοδότηση αυτής της ανθρωπιστικής ε, αντιμετώπισης θα καλύψουμε τις πιο βασικές και πιο επίγουσες ανάγκες που έχουν οι Ιρακινοί οι ίδιοι. Για να μπορέσουμε να έχουμε να σας πούμε καλύτερα και πιο ευχάριστα πράγματα και ειδήσει για τα δεινά αυτή τη φρικτή τραγωδία των Ιρακινών. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στο Γιάνν Έγκελαντ που είναι Γενικός Γραμματέας ε, του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω με συγχαρητήρια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τη διοργάνωση αυτής της διάσκεψης. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η καιρή και πάρα πολύ επίκαιρο αυτό για τους αμάχους του Ιράκ. Χαίρομαι ε, που βρίσκομαι στο ίδιο πάνελ με συναδέλφους από τον ΟΗΕ και την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Εκπροσωπώ μία από τις πολλές ΜΚΟ ε, και οργανώσεις ε, Ιρακινές που σήμερα δραστηριοποιούνται επί τόπου. Έχουμε ε, χιλιάδες εργαζομένους επιτόπου. Πολλά κάνουμε, μπορούμε ακόμα περισσότερα με τη δική σας βοήθεια. Έχουμε τρεις παράλληλες κρίσεις που εξελίσσονται και ε, επιδεινώνονται ταυτόχρονα. Είναι η κρίση της προστασίας που σημαίνει είναι τεράστια η βία και κλιμακούμενη εις βάρος των αμάχων. Είναι αρχαίες κοινότητες, μειονότητες, θρησκείες, οι οποίες σπαράζονται και ε, διαχωρίζονται και διασκορπίζονται ανά το Ιράκ αλλά και ανά την Ιφίλιο. Κοινότητες και πολιτισμοί που ε, ζουν εκεί ε, εδώ και χιλιάδες χρόνια και τώρα καταλήγουν στις πιο ελεηνές συνθήκες. Και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ανεπανόρθωτο. Και αυτή τη στιγμή που συζητούμε ένοπλοι σκοτώνουν, τραυματίζουν, βιάζουν, κακοποιούν ε, γυναίκες και παιδιά ε, σε καθεστώς πλήρης ατιμορρησίας. Και βλέπουμε ως ανθρωπιστικές οργανώσεις ότι υπάρχει και άλλη κρίση που βαθαίνει, που είναι η κρίση πρόσβασης εκεί. Γιατί υπάρχει μια εμπλοκή, ε, επίθεση σε ανθρωπιστική βοήθεια και δεν τους αφήνουν οι ένοπλοι ε, τους αμάχους να ξεφύγουν, να σώσουν τη ζωή τους ή να φτάσουν στα δικά μας καταφύγια. Ας πούμε, στην επαρχία Ανμπάρ σήμερα βλέπουμε ανίποτη ε, συμφορά. Σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες, μάλλον εκατό χιλιάδες αναγκάστηκαν να φύγουν τις τελευταίες μέρες. 85% σχεδόν όλοι δηλαδή. Τώρα δεν είναι σε θέση να ξεφύγουν ε, από τα πεδία των μαχών ή από τις περιοχές της ένοπλης σύραξης. Και είναι και πολύ δύσκολο να φτάσουμε εμείς σε αυτούς. Είναι κλειστές οι γέφυρες, είναι κλειστοί οι δρόμοι που βρίσκουν μπροστά τους και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Ποια είναι λοιπόν η πικρή πραγματικότητα. Σε πάρα πολλά σημεία δεν μπορούν οι άμαχοι να ξεφύγουν από εκεί που είναι για να φτάσουν στη δική μας βοήθεια και εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε σε εκείνους. Αυτό θα πρέπει να τερματιστεί δεν μπορεί. Δεν είναι τσουνάμι. Είναι ανθρωπογενής η κρίση. Δεν είναι καμιά θεομηνία. Μπορεί να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Η τρίτη κρίση είναι η κρίση της ε, παροχής βοήθειας. Και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη των χρημάτων. Η χρηματοδότηση ούτε κατά διάνοια δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις τρομακτικές ανάγκες εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι στο χείλος του γκρεμού κυριολεκτικά ήταν πολύ γενναιόδορες οι ίδιες οι Ιρακινές κοινότητες, ο πληθυσμός. Έχουν ε, αγκαλιάσει τους ε, εκτοπισμένους που μπορεί να είναι μακρινοί συγγενείς, δεν είναι τέλειως άγνωστοι. Η κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση ήταν πάρα πολύ γενναιόδορη γιατί δέχεται στους κόλπους τους ε, και Σύρους και άλλους Ιρακινούς και τώρα θα πρέπει οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, οι Ασιάτες και οι Αραβικές χώρες να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Εμείς, ε, ανθρωπιστικές ΜΚΟ, έχουμε πολλούς εργαζομένους επιτόπου σε πολλά σημεία και ζητούμε ε, πλήρη και ταχεία ε, χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου που μόλις μας παρουσίασε η Λις Γκράντε. Θα πρέπει να έχουμε πλήρη χρηματοδότηση, είμαστε εταίροι, βεβαίως πολλοί από εμά έχουμε και άλλες ανάγκες ε, και άλλες εκκλήσεις πέρα από αυτή την κοινή μας έκκληση. Τέλος. Καταλαβαίνετε ότι η ανθρωπιστική κρίση ανακουφίζει μόνο, δεν τερματίζει αυτό τον πόνο. Καλούνται τώρα οι ηγεσίε στο Ιράκ, πολιτικέ, θρησκευτικέ και πολιτισμικέ, να καθίσουν κάτω σε ένα τραπέζι και να συζητούν μεταξύ του και με του εκπροσώπου των μειονοτήτων για να κάνουν ειρηνικές πολιτικές συμφωνίες. Είναι ο μόνος τρόπος. Οι περιφερειακές και διεθνείς δυνάμεις θα πρέπει να σταματήσουν τις αντιπαλότητες και τους διαξυφισμούς τους που προκαλούν ανίποτα δεινά πόνο δίνει για τους Ιρακινούς. Θα πρέπει να ε, οθήσουν με συνοχή όλα τα μέρη για να βρεθεί κάποια λύση στο Ιράκ και για το Ιράκ. Εμείς είμαστε μερόληπτοι, ανεξάρτητοι ως ανθρωπιστική βοήθεια και διεπόμεθα από την αρχή της ουδετερότητας ε, στις πολιτικές συγκρούσεις και στις θρησκευτικέ διαμάχες. Δεν παίρνουμε το μέρος καθενός. Πηγαίνουμε σε όποιον έχει ανάγκη, ανεξαρτήτως ποιος ελέγχει την περιοχή αυτή και ποιοι είναι οι πραγματικοί κυρίαρχοι. Η αντιτρομοκρατική νομοθεσία δεν θα πρέπει να μας εμποδίζει να φτάνουμε εμείς τα θύματα της τρομοκρατίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουν αυτό οι βουλευτές. Ε, δεν θα πρέπει να έχουμε παράπλευρες συνέπειες ή ανεπιθύμητες συνέπειες και παρενέργειες για να μην μπορούμε να βοηθούμε τα θύματα. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα, περισσότερα χρήματα, περισσότερη πρόσβαση, περισσότερη ασφάλεια και περισσότερη προστασία για αυτούς που βοηθούμε. Οι δικοί μας εργαζόμενοι επιτόπου έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση και προσβλέπουν στο αποτέλεσμά της. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Μπάρμπαρα Νοσόθη που είναι ε, αναπληρώτρια ε, γενική εκτελεστική συγγνώμη, διευθύντρια του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος. Ευχαριστώ. Είναι τιμή για μένα να σας μιλάω σήμερα σαν εκπρόσωπος της Παγκόσμιου Οργάνωσης για, τα, για την παροχή επιστημικής βοήθειας και να απευθύνω έκκληση όσον αφορά το θέμα του Ιράκ, εκ μέρους του Ιράκ. Να ξεκινήσω ότι το παγκόσμιο αυτό πρόγραμμα για τη διατροφή πιστεύει ότι η πρόσβαση στο, στο σωστά τρόφιμα είναι ακρογωνίως λήθος για ισότιμη, δί, ισότιμο δίκαιο και κόσμο που ευημερεί. Η ασφάλεια τροφίμων συμβάλλει στην φυσική ασφάλεια και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα εκ μέρους όλων των οργανισμών να απευθύνουμε έκκληση για στήριξη. Το παγκόσμιο αυτό πρόγραμμα για τη διατροφή προσπαθεί να καταπολεμήσει την πείνα στο Ιράκ από το 1991, να παράσχουμε τρόφιμα σε κόσμο τον οποίον είχε διακοπεί η ζωή τους από φυσικές καταστροφές και από σύγκρουση. Ήταν μια χώρα πλούσια σε πετρέλαιο, αλλά η ανάπτυξη του Ιράκ εμποδίστηκε λόγω συνεχών σειράξεων. Η προστασία των πλέον ευάλωτων Ιρακινών και των φτωχότερων και των οικογενειών που εξαρτώνται από εξαρτώνται από τη, τα αποτελέσματα των βιοπραγιών είναι μια πρόκληση. Το 2012 το Ιράκ άνοιξε τα σύνορά τους προς τα πρόσφυγες από τη Συρία και στις βόρειες και στις δυτικές επαρχίες και, θέλαμε, και δώσαμε τρόφιμα στους πρόσφυγες, στους Σύρους το 2014 όταν έγιναν και πρόσφατες ε, συγκρούσεις εκεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτής που έδωσαν 10 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα μας για το φύτο 2014 για να βοηθήσει τους εκτοπιστέντες Ιρακινούς και 4 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τους ε, Σύρους πρόσφυγες στο Ιράκ. Αυτά τα χρήματα μας βοήθησαν να αγοράσουμε 10.000 μετρικούς τόνους ε, δεμάτων με τρόφιμα για τις οικογένειες για να θρέψουμε 750.000 Ιρακινούς που είχαν ανάγκη και να δώσουμε πάνω από 3,5 εκατομμύρια δολάρια σε δετία και ε, πάρα πολλά δέματα με τρόφιμα για περίπου 150.000 Σύρους πρόσφυγες στο βόρειο τμήμα της ε, χώρας. Η κατάσταση όμως επιδεινώνεται όπως γνωρίζουμε όλοι. Στην αρχή του 2014 στο Ανμπάρ ξέσπασαν οι μάχες και αυτό οδήγησε στο να έχουμε εσωτερικού εκτοπιστέντες. Ε, πλήγησαν οι Ρακίνοι από τον Ιανουάριο και μετά από την Ευρωπαϊκή. Λοιπόν, κινητοποιηθήκαμε γρήγορα και βοηθήσαμε τους εκτοπιστέντες διότι αυτοί επιδίκουν να βρουν ασφάλεια ε, όσο ήταν εκτοπιστέντες. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Ιούνιο του 2014 όταν κατακτήθη η Μοσούλη και άλλες μεγάλες πόλεις στις βόρειες και κεντρικές περιοχές. Οι οικογένειες υποχρεώθηκαν να ξεφεύγουν και να πηγαίνουν από περιοχή και περιοχή και αναπτύσσαμε ειδικό πακέτο ε, διαφόρων ε, τροφίμων, ειδικά για το Ιράκ, έτοιμων τροφίμων, ε, και με δαμάσκηνα και άλλα τρόφιμα. Στην Ινεβή και στη Σύντρα άρχισαν να ξεφεύγει ο πληθυσμό προ τα βόρεια και εμεί ανοίξαμε ε, κουζίνες που έδιναν ε, δύο γεύματα ζεστά ε, γεύματα καθημερινά σε 224.000 ανθρώπους, ανθρώπους που έχασαν ε, τα πράγματά τους, τις, τους φίλους τους, τα σπίτια τους και καταβάλαμε προσπάθειες, ακούγαμε τις πληγήσεις ε, κοινότητες ε, μέσω διαβουλεύσεων που είχαμε οργανώσει. Πήραμε τις πληροφορίες, χρησιμοποίησαμε για να βελτιώσουμε τον προγραμματισμό, να αλλάξουμε τα καλάθια με τα τρόφιμα και να καλύψουμε καλύτερα τις ανάγκες των παραληπτών. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει σωστή παρέμβαση που απευθύνεται στους σωστούς ανθρώπους, σωστή στιγμή, με το σωστό τρόπο. Ξεκινήσαμε να παρέχουμε λοιπόν δελτία τροφίμων σε αστικές περιοχές των κουρδικών περιοχών. Πέρσι τον ε, Νοέμβριο δώσαμε στους πιστέντες Ιρακινούς οικογένειές τους δυνατότητα να επιλέξουν τη δική τους διατροφή. Εξ, εξαργύρωνα σε τοπικά καταστήματα αυτά τα δελτία αγοράσουν αυγά, γάλα, τυρί, κοτόπουλα, οποροκυπευτικά μεταξύ άλλων προϊόντων. Περίπου 470.000 ανθρώπων παίρνουν αυτά τα δελτία τα μηνύα. Δηλαδή δίνουμε περίπου 7 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια που ε, δίνουμε στην τοπική κοινωνία στις κουρδικές περιοχές. Οι συγκρούσεις τελευταίο δίμηνο συνέχισαν να δημιουργούν νέους εκτοπιστέντες. Στην Ανμπάρ περίπου 200.000 άνθρωποι ε, έφυγαν από το Ραμάντι. Ε, συνεργαστήκαμε στενά με άλλες υπηρεσίες, με τη UNICEF και άλλους διεθνείς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, βοηθώντας τον κόσμο με τρόφιμα έτοιμα να φαγωθούν και διάφο... νερό και διάφορα πακέτα με προϊόντα υγιεινής όταν κατέφθαναν στους καταβλισμούς στα σημεία ελέγχου. Έγινε κοινή προσπάθεια και εμείς δώσαμε τρόφιμα, διανύμαμε τρόφιμα σε περίπου 210.000 ε, ανθρώπους Όλη η μέρα εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε στους επιθέντες Ιρακινούς και εξακολουθήσαμε να προστατεύουμε και τους ευάλωτους Σύρους. Τους δίναμε επιστηστική βοήθεια και δελτία τροφίμων και το 2015 με παρκή στήριξη θέλουμε να κλιμακώσουμε την επιχείρησή μας ούτω ώστε να βοηθήσουμε τους καταβλισμούς των Σύρων όπου υπάρχει δυνατότητα να βοηθήσουμε και το λιανεμπόριο έτσι μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε τρόφιμα αλλά να έχει και επιλογή. Δυστυχώς η χρηματοδότηση άρχισε να μειώνεται. Λείπουν χρήματα και αρχίσαμε να περικόπτουμε την ενίσχυση που δίνουμε στους Σύρους και τους Ιρακινούς πρόσφυγες. Αυτοί που ζουν στους καταβλισμούς είναι λιγότερο να έχουν δουλειές από εκείνους που ζουν με φίλους και οικογένειες ή στα σχολεία ή στα τζαμιά και έπρεπε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις για να προστατεύσουμε τους πλέον ευάλωτες. Οι εκτοπιστέντες Ιρακινοί που ζουν σε καταβλισμούς εξακολουθούν να παίρνουν αυτά τα δελτία για τα τρόφιμα, αλλά έπρεπε να μείνουμε μειωμένα πακέτα σε εκείνους που ζουν εκτός καταβλισμών. Περικόψαμε και την τιμή των δελτίων από 26 δολάρια στα 16 δολάρια Αμερικής. Επίσης όλο και περισσότερο βάζουμε προτεραιότητα για τα μυστική βοήθεια προς πλέον ευάλωτους Σύρους πρόσφυγες οικογένεια σα και μειώνουμε τα επίπεδα τη βοήθεια για του άλλου. Βεβαίω αυτά τα ενημερώνουμε τον κόσμο πριν κάνουμε τη διανομή για αυτές τις αλλαγές. Αυτή η μείωση της βοηθείας έχετε μια εποχή όπου η ασφάλεια των τροφίμων μειούται. Χρησιμοποιούμε ε, έλεγχο για να έχουμε εικόνα όσον αφορά την κατάσταση της ασφαλείας, ασφαλείου εφοδιασμού ΡΑΚ. Τον Απρίλιο οι μάχες των Μπαρ οδήγησαν αύξηση των τροφίμων, τιμών των τροφίμων κατά 28% στην σύγκριση με τον ε, Μάρτιο και τα ημερομίστια μειώθηκαν. Ε, κάναμε μαζί με τον ΦΑΟ έρευνε. Ξέρουμε ότι 25% του κόσμου δεν έχει επαρκή αγοραστική δύναμη, οπότε του λείπουν γεύματα ή τρώνε λιγότερα από την ημερήσιε απαιτήσει, όσον αφορά τη δοσολογία. Και άλλε επαρχίε δεν πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Ανησυχούμε πάρα πολύ, διότι περαιτέρω μείωση της επισητιστικής βοήθειας θα επιδεινώσει την κατάσταση και έτσι απευθύνουμε και εμείς έκκληση για τα 180 εκατομμύρια δολάρια. Χρειάζεται κατεπηγόντας χρήματα αγοράσουμε τρόφιμα και δελτία που θα βελτιώσουν την ασφάλεια τροφίμων όσον αφορά τους εκτοπιστέντες ήρους και ρακινούς για το υπόλοιπο έτος. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου κλείνοντας να πω το εξή. Αναγνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και το κόστος της αδράνειας θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος της δράσης. Σας απευθύνω έκκληση, σας ζητώ τη στήριξή σας και σας ευχαριστώ για το έργο που έχετε επιτελέσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πατρίκ Ιουσέφ που είναι επικεφαλής ε, του Γραφείου της Βαγδάτης του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Κυρίε και κύριοι Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που προσκαλέσατε τη Διεθνή Επιτροπή του ε, Ερυθρού Σταυρού σε αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση και στο πάνελ αυτό συγκεκριμένα. Βλέπετε πόσο βαθιές σχέσεις έχουμε, αλλά τονίζω ότι και βασικά χαρακτηριστικά της δουλειάς μας, ε, συντονισμός επιτόπου ανάμεσα στον ΟΗΕ, τη Διεθνή Κοινότητα του Ερυθρού Σταυρού, τους ε, τοπικούς φορείς, ε, της διεθνής ε, ΜΚΟ αλλά και ε, τους Ιρακινούς θεσμούς. Έχουμε κοινέ αξίες και αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε μια ευρύτερη οικογένεια. Νομίζω ότι οφείλουμε να προσέξουμε και να δώσουμε την δέουσα σημασία στο πεπρωμένο του Ιρακινού λαού. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα που ε, εδώ και πάνω από 13 χρόνια πλήττεται από αυτή την καταστροφή εδώ και 30 χρόνια πλήττεται από την κρίση. Ε, και παρά την ε, εσωτερική αλληλεγγύη που βλέπουμε σε ολόκληρη τη χώρα διαπιστώνουμε ότι ε, βρέχει μακροπρόθεσμα, έχουμε σοβαρούς αντικτύπους για πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και πραγματικά πιστέψτε με πρόκειται για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις διότι ασχολούμαστε με περιστατικά που ποτέ ανθρώπων που ποτέ δεν έλαβαν αποζημίωση που κανείς από τον πόλεμο Ιράκ-Ιράν ή από τον πόλεμο Ιράκ ε, ε, Κουβέιτ ε, δεν τους έψαξε κανείς ε, και με την τωρινή διαμάχη απλώς ε, οι ανάγκες. Δεν χρειάζεται τώρα να επαναλάβω όλα αυτά που μας είπε Λίζε. Μας μίλησε για 2,8 εκατομμύρια. Νόμιζα ότι είχαμε σταματήσει αυτό. Τώρα έχουμε ανέβει στο 2,9. Κάθε εβδομάδα βλέπουμε νέα ανησυχητικά νούμερα στέγη, ιατρική περίθαλψη, ανάγκη σε τρόφιμα αυξάνονται καθημερινά και κυρίως δοκιμάζονται οι δοκιμάζεται το δυναμικό ε, πεπειραμένων οργανώσεων, ανθρωπιστικών οργανώσεων με τις αυξημένες αυτές ανάγκες. Συνεχίζονται οι πολεμικές σειράξεις σε όλες αυτές τις περιοχές και χάνεται η ελπίδα ε, για έγκαιρη παρέμβαση. Ταυτόχρονα ο επειδή πολύ μεγάλα τμήματα του πληθυσμού βρίσκονται σε περιοχές μπόλεμες που δεν ελέγχει η κυβέρνηση, ε, δεν υπάρχει καμία πρόσβαση και δεν έχουμε στοιχεία για αυτούς. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρέμβασή σας ε, στον τομέα αυτό, διότι ε, οι διεθνείς θεσμοί ε, του, του Ιράκ καθώς και η διεθνής κοινότητα του Ερυθρού Σταυρού μπορούν ε, να δώσουν βοήθεια διασχίζοντας ε, και σύνορα. Στην Ελχαμπανίλια την τουριστική πόλη, έχουμε μοιράσει παραδείγματο χάρη νερό, τρόφιμα και αυτό που μας σώκαρε περισσότερο είναι όταν μας φώναζαν οι άνθρωποι και μας λέγανε τραβήξτε βίντεο, πάρτε φωτογραφίες ούτως ώστε να δείξετε ότι ε, χρειάζονται προστασία γιατί μπορεί και να εκτοπιστούν και πάλι και να χαθούν μετά, να μην, να μην ξέρει κανείς που είναι και έτσι τεκμηριώνει τη ανάγκη για προστασία, χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος όπου μπορεί να νιώθει ασφάλεια η οικογένειά τους. Και για να μην υπάρχει καμία παρανόηση θα ήθελα να σας πω ότι κατά τη γνώμη, κατά τη γνώμη της οργάνωσής μου ανεξαρτήτως πολιτικού βάρους ε, και με ενιών όπως ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, και τα το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ανθρωπιστική δράση, οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, η ύψη σημασία πρέπει να αποδοθεί στην νομική ταξινόμηση της κατάστασης. Πέρσι κατατάχθηκε στην κατηγορία των ενόπλων σειράξεων του Ιράκ διεθνώς αναγνωρισμένη κατάταξη από την κυβέρνηση του Ιράκ βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και δυνάμει των συνθήκων της Γενέβης. Εάν αποκλίνουμε από την εφαρμοσιμότητα και την ανάγκη συμμόρφωσης με τις αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου επί το που σίγουρα θα είναι επιζήμια για αυτούς που υποτίθεται ότι χρήζουν προστασίας ε, βάσει του δικαίου. Και όσοι δεν ε, συμμετέχουν πλέον σε εχθροπραξίες κυρίως. Αυτοί που δεν ενεργοποιούνται πλέον στρατιωτικά θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχουν ε, οι καλοί και οι κακοί πολίτες, ε, τρομοκράτες και μη τρομοκράτες. Ε, προστατεύονται όλοι από το διεθνές δίκαιο και είτε μας αρέσει είτε όχι όλοι χρήζουν προστασίας. Εν συνόψη, υπάρχουν οι εξή ε, τάσει στο Ιράκ. Ε, σε πυκνοκατοικημένε ε, περιοχέ κλιμακώνονται οι εντάσει και οι σειράξει. Πολύ ανησυχητικό αυτό γιατί αυξάνει το αριθμό των θυμάτων στον πληθυσμό. Όπω είπε και η Δόκτωρ Καν, σε σχέση με τις ιατρικές επιχειρήσεις και την προστασία των ιατρικών καταστάσεων και εγκαταστάσεων παροχής ε, ε, ιατρικών ε, υπηρεσιών θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχιση των δράσεων. Υπάρχουν και αυτοί οι όμοιροι που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους και ε, δεν θέλω να υπονομεύσω τη δυνατότητα ε, της Ιρακινής ε, κυβέρνησης να συλλαμβάνει και να δρά και να παίρνει εχμαλό τους, αλλά για αυτούς τους κρατούμενους θα πρέπει να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής μεταχείριση. Επίσης, η εξαφανισμένη και τώρα επιστρέφω ε, ε, επιστρέφω στην αρχική της παρέμβασής μου ο αυξημένος αριθμός αγνωμένων ε, στον ε, κόσμο είναι το Ιράκ τα τελευταία 30 χρόνια και η αγωνία των οικογενειών εδώ ασχολούμαι περισσότερο με τις οικογένειες αλλά πέραν αυτού σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και την Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και τη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου προσπαθούμε να ξεθάψουμε και συλλογικούς τάφους να βρούμε πού βρίσκονται αυτοί οι αγνοούμενοι. Πέρα από το τις πρωτοβουλίες, τα κουτιά πρώτης βοήθειας, την ε, ορθοπαιδική και ε, αποκατάσταση, ε, φυσιοθεραπείες, δράσεις ε, παροχή τροφίμων και ποσίμου νερού, ε, σε διάλογος με την Ιρακινή Βουλή, με τα Υπουργεία, την κυβέρνηση αλλά και όλους όσους ε, εμπλέκονται επί τόπου. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα δράση, πηγαίνουμε σε κέντρα κράτησης, παραδείγματος χάρη, και βλέπουμε ότι ε, ότι φτάνουν στους 35-40 χιλιάδες. Το βάση των συνδικών της ε, Γενέβης ε, και του άρθρου 1 συγκεκριμένα όλοι θα πρέπει πέρα από το Ιράκ να φροντίσουν ούτως ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με το διεθνές δικαίωμα, με την κατάρτιση, με την αρρωγή, με την το να βοηθήσουν το Ιράκ να καταλάβει τι διακυβεύεται για το ίδιο το κράτος και για την ιστορία και για την περιοχή. Ε, για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για το Ιράκ θα πρέπει σε αυτή τη μεταβατική περίοδο να φροντίσουμε να εφαρμοστεί ε, σωστά το δίκαιο ούτω ώστε να υπάρξει συμφιλίωση, σταθεροποίηση και αποκατάσταση ναι, μεν, αλλά το πιο σημαντικό είναι να, γίνει αυτό για τα θύματα του πολέμου, της ε, ε και ε, νομίζω ότι πρόκειται για κοινή μας υποχρέωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ιουσέφ. Θα αρχίσει η συζήτηση. Ε, ε, θα ήθελα προηγουμένως όμως να δώσω το λόγο στον κύριο Λισίντη που είναι υπουργό Προγραμματισμού της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Shall I speak from here? Θα μιλήσω από εδώ. Excellencies. Χαίρετε. Εξοχότητες, κύριε Πρόεδρε της Ιρακινής Βουλής, κύριε Πρόεδρε Μπροκ, κυρία Μακάβαν, κύριε Πίτρο Στυλιανίδη, Δόκτωρ Τόνι Λέικ, Δόκτωρ Τσάνκ, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και τα Ηνωμένα Έθνη για την διοργάνωση αυτής της τόσο επίκαιρης συνεδρίασης. Μας περιβάλλουν σύραξη, βία και ριζοσπαστικοποίηση. Εκτιμώ πάρα πολύ ε, τη δυνατότητα που μας παρέχει να μιλήσουμε. Ανησυχούμε πάρα πολύ από το Ιρακινό Κουρδιστάν. Ε, Μην μείνουμε στο περιθώριο από τις ε, διεθνείς συζητήσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εμείς έχουμε τους Πεσμεργά εκεί που μάχονται επί τόπου σε ένα μέτωπο που είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα η γραμμή του μετώπου. Πάνω από 1.300 Πεσμεργά έχουμε θύματα και πάνω από 6.000 τραυματίες από την αρχή της σύγκρουσης αυτής. Και θα ήθελα εδώ να ζητήσω τη βοήθεια των μεμονωμένων κρατών μελών να βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν οι τραυματίες Πεσμεργά. Εκπροσωπούμε την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, του Ιράκ και υποστηρίζουμε την έκκληση του ΟΗΕ για να χρηματοδοτηθεί το ανθρωπιστικό σχέδιο για όλο το Ιράκ. Πολλές περιοχές του Ιράκ είναι σήμερα σε αποσταθεροποίηση, αλλά εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στη δική μας περιφέρεια, διότι εκπροσωπώ την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν. Ο λαός και η κυβέρνηση της περιφέρειας του Κουρδιστάν τώρα είναι στο μέτωπο και του πολέμου και της ειρήνης ταυτόχρονα και ο λαό και η κυβέρνηση του Κουρδιστάν στο Ιράκ. Πολεμούμε με τις δυνάμεις του ISIS και ε, οικοδομούμε την ειρήνη δεχόμενη μεγάλους αριθμούς σύρων προσφύγων και Ιρακινών εσωτερικά ε, εκτοπισμένο Από το 2005 και μετά έχουν αρχίσει οι Ιρακινοί να διαφεύγουν προς το Κουρδιστάν. Το 2012 το Κουρδιστάν άνοιξε τις σύρες για ε, πρόσφυγες από τη Συρία και διατήρησε ανοιχτές αυτές τις πύλες. Το δεύτερο εξάμεινο του 2014, μέσα σε λίγους μήνες, σχεδόν ένα εκατομμύριο Ιρακινών αδελφών μας, χριστιανών, γεζιντή, Κούρδων, Τουρκομάνων, Αράβων, ε, μπήκαν στην κουρδική περιοχή του Ιράκ. Σήμερα τουλάχιστον ένας στους τέσσερις στο Κουρδιστάν είναι εκτοπισμένος από κάπου αλλού. Σε όλη την επαρχία ο λόγος αυτό είναι ένας προς δύο. Και όσο έρχονται περισσότερο εκτοπισμένοι μειώνεται αυτή η σχέση. Μέχρι τώρα 5 εκατομμύρια φιλοξενούν περίπου 1,7 εκτοπισμένους, Ιρακινούς και Σύρους πρόσφυγες. Και οι δύο κοινότητες πλήττονται και χρειάζονται υποστήριξη. Διεθνώς δεν γίνεται εισήγηση των ε, προσφύγων ε, με τους εσωτερικά εκτοπισμένους ή δεν αναμειγνύονται, αλλά εμείς όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, τις ίδιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι αυτοί, είτε είναι πρόσφυγες είτε είναι εσωτερικά εκτοπιστέντες. Σας παρακαλώ, καθίστε μια στιγμή και αναλογιστείτε όλα αυτά τα νούμερα και σκεφτείτε πώς εσείς θα ανταποκρινόσαστε αν υπήρχε τέτοια ραγδαία αύξηση πληθυσμού τόσο γρήγορα στις δικές σας εκλογικές περιφέρειες. Πάνω από 30 καταβλισμούς έχουμε, Παύλα Πόλης, ε, κατασκευάσει, αλλά αγωνιζόμαστε να βρούμε λεφτά και να ε, τρέξουμε τη λειτουργία. Παρ' όλα αυτά, ε, είναι πολλοί ακόμα εισιτορικά εκτοπισμένοι που ζουν σε εκτρές ε, συνθήκες, σε γιαπιά και σε άλλα κατάλληλα στεγάσματα. Και πολλοί με το καιρό έχουν μετατοπιστεί και ε, παρόλη τη φιλόξενη υποδοχή ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δύο τρίτα των παιδιών των εκτοπισμένων και μισά από τα παιδιά των προσφύγων δεν είναι σε κανένα σχολείο και σε κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα γραμμένα. Δεκάδες χιλιάδες γυναικών και μικρών κοριτσιών κινδυνεύουν όχι να χάσουν τη ζωή τους ε, ε απαραίτητα, αλλά ε, να χάσουν την ευημερία τους. Ε, η φτώχεια έχει υπερδιπλασιαστεί στο Κουρδιστάν, έχει μειωθεί το βιωτικό επίπεδο, η επισητιστική ασφάλεια πλήττεται, η κατάσταση υγείας επιδεινώνεται με απειλές χολέρας να εμφανιστεί το καλοκαίρι σε ορισμένες περιοχές. Και έχουν επίσης διατραχθεί πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Η κατάσταση στο Κουρδιστάν είναι ένα μείγμα επίγουσας ανάγκης και αντίστασης ταυτόχρονα. Η Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει την κοινωνική και πολιτική επίπτωση της κρίσης στο Κουρδιστάν σε μια μελέτη στα τέλη του 2014 και αρχές του 2015. Το ΑΕΠ μειώθηκε από 8% που ήταν το 2013 σε 3% το 2014. Η ανεργία εκτινάχθηκε και γιατί μπαίνουν οι πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένοι στην αγορά εργασίας και ρίχνουν τους μισθούς. Η Τράπεζα Παγκόσμια έχει υπολογίσει ότι το κόστος όλων αυτών είναι τουλάχιστον 1,4 δις ε, δολάρια για το έτος 2015. Το ποσό αυτό είναι σε επιπλέον προϋπολογισμός. Γι' αυτό ε, είμαστε εδώ σήμερα. 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το κόστος σταθεροποίησης για την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν εκτός από τα 500 εκατομμύρια τα οποία ζητεί ε, ο ΙΕ για τη χρηματοδότησή μας. Όπως είπε προηγουμένως η Μπάρμπαρα Νόσγουόρθη, το κόστος της αδράνειας ίσως πραγματικά είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος της δράσης. Τώρα, σκεφτείτε παρακαλώ μια στιγμή τη σχέση μεταξύ σταθεροποίησης ε, μιας εμπόλεμης περιοχής ε, και πώς, πώς συνδέεται αυτό με τη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Σας παρακαλώ να το σκεφτείτε και να δείτε αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει σχέση. Εμείς στο Κουρδιστάν κάναμε ό,τι μπορούμε και ό,τι μπορούσαμε. Και μας αξίζει πραγματικά περισσότερη προσοχή και περισσότερη βάση να δοθεί. Τη στιγμή που η δημοσιονομική μας κατάσταση είναι ήδη δεινή, δεν έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε αυτές τις υποδομές, τους καταβλισμούς ή να δώσουμε αυτό το πλήρες φάσμα ε, δημοσίων υπηρεσιών σε πρόσφυγες που φιλοξενούμε ή σε εσωτερικά εκτοπισμένους. Είναι απλήρωτη η να δωσουμε αυτο το πληρες φασμα υπηρεσιων σε προσφυγες που φιλοξενουμε η σε εσωτερικα εκτοπισμενους ειναι απληρωτη η δημοσια πάλι μας και είπε για τους τελευταίους τρεις μήνες. Καταλαβαίνετε και θα συμφωνήσετε ότι είναι αφόρητη πλέον αυτή η κατάσταση. Ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την οικονομία μας. Το Ιράκ θεωρείται μια χώρα μεσαίου εισοδήματος και επειδή έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου και γίνεται ο πόλεμος ε, το Ισλαμικό κράτος και για πολλού άλλου λόγους είναι πολύ περίπλοκη η οικονομική κατάσταση. Του επόμενου μήνες ο πόλεμος κατά του Ισλαμικού κράτους θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περισσότερες εκτοπίσεις. Αυτή τη στιγμή που σα μιλώ δεν είμαι βέβαιο ότι όλοι είμαστε συλλογικά προετοιμασμένοι να απαντήσουμε σε τέτοιες μετατοπίσεις πληθυσμών Είτε είναι από το Ραμάντι, από τη Μοσούλη ή από αλλού. Ο λαός και η κυβέρνηση του Κουρδιστάν έχουν δείξει φιλοξενία, γενεδορία, ε, μακρόχρονικό διάστημα και έχουν αφήσει ανοιχτές τις θύρες για τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους, αλλά ε, είμαστε σε ένα σημείο καμπής. Ε, χρειαζόμαστε την υποστήριξη και τη διεθνού κοινότητα και των μεμονωμένων κρατών τη ευρωπαϊκή Ένωσης για να χρηματοδοτήσουν την έκκληση του ΟΗΕ και να βοηθήσουν την κυβέρνηση του Κουρδιστάν με ανθρωπιστική βοήθεια και με βοήθεια υποστήριξη της οικονομίας μας. Χωρίς ισχυρή υποστήριξη και διαρκή της διεθνούς κοινότητας αποκλείεται να αντέξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Εδώ στην Επιτροπή μας γίνεται μεγάλος λόγος για τις προσπάθειες ε, του κουρδικού λαού ε, και τους αγώνες που δίνει, όχι μόνο στην υποδοχή προσφύγων, αλλά και στο στρατιωτικό σκέλος και η Πεσμεργά, όπως είπατε, και στο Κομπάνι το είδαμε, όχι μόνο στο Ιράκ. Σας ευχαριστώ. Ε, πριν ε, δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Μπράιν Χάιεφ, που είναι αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ιράκ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω όλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την έκτακτη συνεδρίαση και ήταν καλό να ακούσουμε τις μαρτυρίες για τη φρικτή κατάσταση που αντιμετωπίζει ο λαός του Ιράκ και τις διεθνείς ευθύνες που υπάρχουν και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ευθύνες για επίλυση του προβλήματος και να στηριχθεί ο κόσμος που έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και την τραγωδία αυτή και επί σειρά ετών. Θα ξεκινήσω απηχώντας κάποια από τα αναφερθέντα σχόλια τα σχόλια των συναδέλφων από το Κουρδιστάν. Δύο θέματα θέλω να θίξω. Πρώτον, βλέποντας τον αριθμό των εκτοπιστέντων που φιλοξενούνται στο Κουρδιστάν και το πολύ μεγάλο βάρος που αυτό θέτει στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται, υπέχουμε ευθύνη και στο Ιράκ και στο Κουρδιστάν να βοηθήσουμε και την κυβέρνηση και το λαό, διότι είναι πολύ ανοιχτή όσον αφορά τους εκτοπιστέντες που υποδέχονται στην περιοχή. Ε, δεύτερον, έχουμε και άλλη ευθύνη. Και η Βαγδά την ευθύνη, έχει ευθύνη να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις που έδωσε τις οικονομικές όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Η κατάσταση θα βελτιωθεί σημαντικά όσον αφορά τα διπλωματικά ζητήματα αν τελικά τηρηθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Και ε, θα έπρεπε να το πούμε αυτό στη σημερινή συνεδρίαση. Η ανθρωπιστική χρηματοδότηση της οποίας ηγείται ο ΙΕ συμπεριλαμβανομένης αυτής που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα για ανταπόκριση ανθρωπιστική ανάγκη μπορεί να είναι φορέας όχι μόνο για κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και μεγαλύτερη αύξηση της σταθερότητας στην περιοχή και έτσι να βοηθηθεί μια εθνική συμφιλίωση στο Ιράκ. Κάτι που στηρίζουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη αντιπροσωπείας μας μάλλον, καλώντας τους συχνά ανταγωνιζόμενους φορείς όπως είναι το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία να συγχρηματοδοτήσουν τον ανθρωπιστικό σχεδιασμό του ΟΗΕ και να συμμετάσχουν ενεργά στην εφαρμογή, στο σχεδιασμό και στην ε, υλοποίηση αυτού. Οι τρεις προαναφερθέντες ε, περιφερειακοί φορείς έτσι θα έχουν δυνατότητα να θύσουν ε, γύρω από το ίδιο τραπέζι σε ουδέτερο περιβάλλον και να συνομιλήσουν με άλλους ιδρυτικούς εταίρους όπως εμάς στην Ευρώπη για το πώς μπορεί να υπάρξει στενότερος συντονισμός με την κυβέρνηση του Ιράκ και να καλυφθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες και προτεραιότητες στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαμεσολαβητή στη διαδικασία, μεσάζων. Με τέτοια στρατηγική που θα εμπλέκει και άλλους περιφερειακούς φορείς θα βοηθήσει σημαντικά. Και θα βοηθήσει και τον Ιρακινό Πρωθυπουργό που καταβάλει διπλωματική προσπάθεια για να βελτιώσει τη σχέση του Ιράκ με τους περιφερειακούς γείτονες, τους άμεσους γείτονες του Ιράκ. Εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε στη βελτίωση της ποιότητας των προσπαθειών. Ερώτησή μου προς το πάνελ. Σε ποιο βαθμό η Τουρκία, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου έχουν συμμετάσχει στον καθορισμό του αναθεωρημένου σχεδίου για την ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ. Σε ποιο βαθμό συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό Οικονομικά, σε ποιο βαθμό συμβάλλουν σε αυτή τη φάση, είναι πλούσιες χώρες. Έχουν τη δυνατότητα να κωδικοποιήσουν προγράμματα και δράσεις που απορρέουν από το σχεδιασμό σε συντονισμό με την κυβέρνηση του Ιράκ. Αν όχι, τι δυνατότητες υπάρχουν. Μπορεί να εγκαινιαστεί μια νέα εποχή συνεργασίας σαν συνέπεια του ανθρωπιστικού σχεδιασμού που θέλουμε να ετοιμάσουμε. Θέλουμε οι περιφερειακοί φορείς της περιοχής να σπηρίξουν την προσπάθεια. Έτσι θα βοηθηθεί και η ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και η όλη προσπάθεια συμφιλίωσης της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκόμες παρακαλώ. Thank you. I also am grateful. Ευχαριστώ και εγώ είμαι ευγνώμη για, ε, για το σημερινό πάνελ για την ανθρωπιστική ε, δράση. Ο στόχος είναι η εξασφάλιση χρηματοοικονομικής υποστήριξης και εγώ φυσικά είμαι υπέρ. Όμως πρέπει να πούμε ταυτόχρονα ότι Κάνουμε λάθος ε, που εξετάζουμε μόνο την ανθρωπιστική διάσταση εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζουμε ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τις αυθύνες μας ε, προβάλλοντας αυτή την ανθρωπιστική δράση. Καλό είναι για ε, την, τον αυτοσεβασμό και την αυτοεκτίμησή μας, όμως δεν αρκεί. Γιατί για τη δράση και την έλλειψη δράσης επίσης φέρουμε ευθύνη. Ε, θα ήθελα λοιπόν, ε, όπως είπε και ο κύριος Τέρκ, ε, να τονίσω και εγώ ότι υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη προς τον Ιρακινό λαό. Το είδα αυτό, η διεισόμαση, από, πήγα από το Ερμπίλ μέχρι το Τεχούκ και επισκέφθηκα καταβλισμούς προσφύγων τον Ιανουάριο και την είδα, την είδα έμπρακτα αυτή την αλληλεγγύη και είναι καταπληκτικό. Και πραγματικά ραγίζει η καρδιά μου όταν βλέπω ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν καταλαβαίνουν Περζίνος πρόκειται και τι διακυβεύεται όχι μόνο για τους Ιρακινούς αλλά και πώς εκείνοι αγωνίζονται για τη δική μας ασφάλεια, γιατί ε, είναι στην πρώτη γραμμή στο, του αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο Ιράκ, όπως και στη Δαμασκό, στη Συρία και ε, επίσης ε, για ε, τα έχουμε κάνει χάλια και στη, στο Ιράκ και στη Συρία. Εμείς ευθυνόμαστε. Ε, πήγαμε εκεί με άλλους τρεις ευρωβουλευτές και επίσης γράψαμε συνέχεια μία επιστολή προς την κυρία Μογκερίνη για να τονίσουμε ότι ακόμη και στο ανθρωπιστικό πεδίο πολλά πρέπει να γίνουν ε, ακόμη και με ταράσει ε, το ότι έχουν κλείσει τα σχολεία στους καταβλισμούς ε, διότι οι Ιρακινές αρχές δεν έχουν πλέον δυνατότητα να τα στηρίξουν χιλιάδες ε, παιδιά, χιλιάδες παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο και τι κάνουμε, κατασκευάζουμε τρομοκράτες έτσι. Τι κάνουμε λοιπόν στην ανθρωπιστική μας ε, δράση. Δεν φροντίζουμε για τα σχολεία και αυτό οφείλεται ε, στην έλλειψη συντονισμού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα στην ΕΧΟ και τα κράτη-μέλη. Ε, είμαστε εκεί αλλά δεν υπάρχει συντονισμός και είναι σοβαρό το πρόβλημα και το υποδείξαμε και στην κυρία Μογκερίνη και στον Επίτροπο Στυλιανίδη. Ελπίζω να, έχει, να υπάρχει τώρα κάπως καλύτερος συντονισμός σε επίπεδο συναρμοδίων επιτρόπων. Επίσης υπάρχουν πολλοί καταβλισμοί άτυποι για τους εσωτερικά εκτοπιστέντε. Αυτό τι σημαίνει, δεν φτάνουν τα λεφτά για όλους και είναι παραπονιούνται και για βασικά πράγματα, έτσι, καθαρό πόσιμο νερό, τρόφιμα και οι μεν, αυτοί που είναι στους άτυπους καταβλισμούς είναι δίπλα στους άλλους, στους επίσημους καταβλισμούς. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Για ε, τις απαγωγές τώρα για τα κορίτσια και για τα παιδιά που έχουν απαχθεί, ε, δεν έχω δει τίποτα, καμία σοβαρή προσπάθεια να γίνεται με τοπικά δίκτυα, με δράσεις τη ε, Ιρακινής κυβέρνησης ε, γίνονται υποτίθεται κάποιε προσπάθειε, όμως εμεί δεν του ε, στηρίζουμε και θέλω να σας ρωτήσω, δεν υπάρχει διεθνής βοήθεια, δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα, διότι αυτοί που ξεφεύγουν τελικά όπως τα κορίτσια ΣΥΝΤΗ, ε, μπορούν να μας δώσουν ε, χρήσιμες πληροφορίες. Ε, ακόμη και από πολιτική σκοπιά δηλαδή είναι σημαντικό να κινηθούμε και να δραστηριοποιηθούμε μέσω ενός τέτοιου προγράμματος. Επίσης, με σοκάρι που δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα. Για να βοηθήσουμε, δεν μιλάμε μόνο για τους μαχητές πεσμέργα που χρειάζονται ειδική ιατρική περίθαλψη. Αυτά τα κορίτσια έχουν τραυματιστεί για ολόκληρη τη ζωή, μα είναι απαράδεκτο, σκανδαλώδες, που δεν έχουμε ένα πρόγραμμα για να τους βοηθήσουμε, διότι αυτά τα κορίτσια δεν μπορούν καν να είναι ε, στην, ε, να, γίνουν, να ενσωματωθούν στην κοινότητα στην οποία ανήκουν. Ένα τομέα στον οποίο χρειαζόμαστε συντονισμό είναι η επανεγκατάσταση. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Άλλη Σίντι. Και να κάνουμε τον παραλληλισμό ανάμεσα σε αυτά που συμβαίνουν τώρα στη Μεσόγειο και αυτά που συμβαίνουν στο Ιράκ, είτε μιλάμε για χριστιανούς, για Ιαζίδη, όλοι μας λένε, εμείς με την πρώτη ευκαιρία που θα έχουμε θα έρθουμε στην Ευρώπη. Είναι θέμα χρόνου. Δεν μπορούμε να κάτσουμε εδώ πέρα. Και οι ηγέτες των θρησκευτικών αυτών κοινοτήτων μας λένε «Μα δεν είναι μόνο θέμα επιβίωσης». Είναι θέμα των επιβίωσης των ε, προ-Ισλαμικών πολιτισμών. Ακόμη πιο σημαντικό είναι αυτό από το να τους βοηθήσουμε να επανεγκατασταθούν γιατί είναι και βασικές ανάγκες. Ε, είδα ε, στο Ερμπίλ ε, την, τον καταβλισμό εστερικά εκτοπισμένων στο προάβλιο της εκκλησίας και ακόμη και εκεί υπήρχε πρόβλημα με, την, με τα σχολεία. Πώς μπορεί να φανταστεί κανείς ότι υπάρχει μέλλον αν δεν καλύπτονται βασικές ανάγκες. Κάποια γελία δε προγράμματα κάποιων χωρών, ειδικά προγράμματα λέει μετανάστευσης για τους χριστιανούς. Μα είναι εντελώς αντιπαραγωγικό αυτό. Είναι ακριβώς ε, το αντίθετο από αυτό που μας, είπαν, που μας οι, οι προκαθήμενοι, οι ηγέτες ε, μην τους βγάζετε από το Ιράκ. Φροντίστε ώστε να συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να παραμείνουν στο Ιράκ. Και όταν θα επανεγκατασταθούν πιο μόνιμα ή μπορέσουν να επιστρέψουν στις χώρες τους και έχουν τις διεθνείς εγγυήσεις, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Και αυτό με επαναφέρει στο βασικό μου μήνυμα δεν κάνει όσα θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς ε, την ε, ε, πολιτική βοήθεια ή ακόμη και την στρατιωτική βοήθεια προς τους μαχητές Πεσμέρια. Εγώ σοκάρομαι όταν βλέπω ότι τα εμπλεκόμενα κράτη-μελή και αυτοί που δίνουν τα όπλα στους Κούρδους, ούτε αυτές οι δύο χώρες δεν μπορούν να συντονιστούν μεταξύ τους. Μα είναι γελίο αυτοί που έχουν αναλάβει την εκπαίδευση των δυνάμων ασφαλεία δεν έχουν συντονιστεί μεταξύ του. Δεν ξέρω αν συντονίζονται σε έναν ευρύτερο συνασπισμό του ΟΗΕ. Μεταξύ του πάντω δεν συνεννοούνται. Και ε, αυτό είναι το πρόβλημα και έτσι δεν μπορούμε να ε, υλοποιήσουμε ε, αυτά που επιδιώκουμε. Και μην ξεχνάμε ότι είναι στην πρώτη γραμμή αυτοί οι άνθρωποι και για τη δική μας ασφάλεια και σωστά τα είπε και ο Μάικλ για του, τις γειτονικές χώρες ε, του Ιράκ που ε, πυροδοτούν τις, τρομοκρατικές, ε, ε τις δυνάμεις στο Ιράκ. Θα είναι πολύ αρνητικό αντίκτυπο η δράση τους. Σας ευχαριστούμε κυρία ε, ήθελα να μιλήσω, όχι ως πρόεδρος, αλλά ως βουλευτής της Ενωτικής Αριστεράς. Εγώ πάντα το επαναλαμβάνω δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα σφάλματά μας. Δεν είναι θεομηνία αυτό που συμβαίνει. Είναι εγκληματικές οι ευθύνε και τα σφάλματα. Φυσικά, εγώ δεν υποστηρίζω τον Σαντάμ Χουσέιν, αλλά το φάρμακο ήταν χειρότερο από την αρρώστια. Πρέπει να δούμε τον αριθμό των νεκρών. Και αυτά δεν τα λέω εγώ. Το 2006 υπήρχε μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης Τζόνς Χόφσκισκινς που έλεγε 600.000 είναι οι νεκροί Ιρακινοί και έκανε μια προβολή αργότερα που μιλούσε για πάνω από 1.400.000 νεκρούς. Είχε δίκιο ο υπουργό όταν μίλησε για τα κονδύλια. όταν ε, φύγανε ε, τα λεφτά ε, από το Ανμπάρ, από το Ντεσπερτάρ, που καταπολεμούσαν την Αλκάιτα, και πήγανε τελικά στην έρημο και άρχισαν να συντονίζονται με τους τρομοκράτες. Αυτό ήταν τελείως ανεύθυνο. Και επιπλέον κάνουμε τα ίδια ασφάλματα με την επέμβαση στη Λιβύη. Τι έχουμε τώρα ένα χάος φτιάξαμε, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Τέσσερα εκατομμύρια ήταν οι εκτοπισμένοι στο Ιράκ, δύο εκατομμύρια εσωτερικοί και δύο εκατομμύρια ε, που τους δέχτηκαν στη Συρία και έχω και δικού μου φίλους που έχουν πάει από εκεί στη Συρία και θέλω να ρωτήσω οποιονδήποτε αρμόδιο μπορεί να απαντήσει από τον ΟΗΕ ή τον Ερυθρό Σταυρό. Τι γίνεται με τους δύο εκατομμύρια Ιρακινούς πρόσφυγες που έχει δεχθεί η Συρία. Υπάρχουν επαφές, γιατί εγώ είμαι υπέρ των επαφών με τη Συριακή κυβέρνηση, όπως έχει σήμερα η κατάσταση. Γι' αυτό επενώ και εκθιάζω την πολύ δύσκολη δουλειά που κάνει ο κύριος Δημιστούρα, ο ειδικό απεσταλμένος για να προσπαθεί να φτιάξει κάποιους χώρους ειρήνης. Ίσως έχει έρθει η ώρα να αρχίσουμε να ξέρουμε ποιος είναι ο σημαντικότερος εχθρός μας εκεί. Κυρίες και κύριοι, είναι αυτοί που αυτό αποκαλούνται κακός Ισλαμικό κράτος. Μια τρομοκρατική οργάνωση είναι που θα πρέπει να καταπολεμήσουμε, να πατάξουμε με κάθε μέσο εντός της διεθνούς νομιμότητας. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να δώσω τώρα το λόγο ε, στο κοινό. Ε, τρία λεπτά έκαστο, διότι κάπως πιέζει ο χρόνος. Ο κύριος Εντουάρ Ροτιέ από τους Γιατρούς χωρί Σύνορα. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλου. Είναι πολύ καλό που είμαι σήμερα και έχω τη δυνατότητα εκ μέρου των Ιατρών χωρί Σύνορα να συμμετάσχω στη σημαντική αυτή διάσκεψη. Τα περισσότερα που είχα να υποθούν υπόθηκαν. Αυτά που θέλαμε να πούμε, καλύφθηκαν. Το μόνο που έχω να πω εντάχει είναι να τονίσω ότι βεβαίω η χρηματοδότηση είναι απολύτω αναγκαία αλλά η χρηματοδότηση ε, απαιτείται μόνο αν υπάρχει πρόσβαση. Αυτό που υπόθηκε και θέλω να τονίσω και εγώ είναι η ανάγκη για ασφαλή πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό σημαίνει και πρόσβαση που δεν χρειάζεται αναδιαπραγμάτευση κάθε φορά που θέλουμε να φτάσουμε σε μια νέα απολευθερωθήσα περιοχή. Κάθε προσπάθισμα καταβάλλονται για τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες να μπορούν να προσέρχονται στους ευάλωτους πληθυσμούς. Μπορούν να γίνουν περισσότερα γι' αυτό. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να διαβιβάσουμε. Τα υπόλοιπα σαφέστατα υπόθηκαν. Σας ευχαριστώ ξανά που μας ε, δώσατε αυτή την ευκαιρία να έρθουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλάν Μπόουμαν ε, είναι αναπληρωτής πρέσβης της αποστολής του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους διοργανωτές που εκάλεσαν τον Καναδά να συμμετάσχει στη διεθνή αυτή συνεδρίαση για το Ιράκ. Προβληματιζόμαστε πολύ από την κρίση και είμαστε σημαντικοί συνεισφοροί στην ανθρωπιστική βοήθεια και θέλουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον συνεργαζόμενοι στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ και όλους τους φορείς που εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Είμαστε στις Βρυξέλλες και γι' αυτό υπογραμμίζω ότι ο Καναδάς ενδιαφέρεται στη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και πέραν αυτού είμαστε εταίροι σε πολλά ανθρωπιστικά ζητήματα και θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση και να αυξήσουμε. Ο Καναδάς ανησυχεί πολύ για τη βία στο Ιράκ και για την ανθρωπιστική συνέπεια που έχει αυτό για εκατομμύρια ανθρώπους που πλήττονται από την κρίση. Καταδικάζουμε τη στόχευση ε, ε, θρησκευτικών μηνοτήτων και αμάχων και τη διάπραξη ε, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά ανθρωπότητα όλα τα μέρη στη σύραξη καλούμε να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και καλούμε τις κοινότητες να επιτρέψουν ανεμπόδιστη και ασφαλή πρόσβαση στους ε, αμάχους που ξεφεύγουν από τις περιοχές ε, σύγκρουσης και να επιτρέψουν επίσης και την πρόσβαση ανθρωπιστικών ε, οργανώσεων, όπως είπαν και για τη σύνορα. Η κυβέρνηση του Καναδά θέλει να δώσει ανθρωπιστική ε, βοήθεια, στήριξη που διασώζει ζωές, εκείνους που εμπλέκονται στην ανθρωπιστική κρίση στον Ιράκ. Έχουμε δώσει 107 εκατομμύρια δολάρια ε, για ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρωπιστικούς εταίρους στο Ιράκ που ανταποκρίνονται στην παρούσα κρίση. Από αυτό το ποσό 80 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν από την αρχή του νεστό έτος. 40 εκατομμύρια από αυτά δόθηκαν σε ανταπόκριση στις προτεραιότητες Fast Track για το Ιράκ που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2015. Ο Καναδά είναι να αντιμετωπίσει τι μακροπρόθεσμε ανάγκε του Καναδά πέρα από τι άμεσε ανθρωπιστικέ ανάγκε και την κρίση. Άλλα 23 εκατομμύρια πρόσφατα ανακοινώθηκαν για αναπτυξιακή βοήθεια και προγραμματισμό θα βελτιώσουν την πρόσβαση υπηρεσίε και θα ενισχύσουν την αντοχή των κοινοτήτων και των κυβερνητικών θεσμών. Τι το τρόπο, η δυνατότητα να ανταποκριθούν οι ανάγκε του πληθυσμού με έναν ολιστικό τρόπο θα ενισχυθούν και τώρα και στο μέλλον. Η καναδική ανθρωπιστική βοήθεια και η σχετική χρηματοδότηση στηρίζει την παροχή τροφίμων, καθαρού νερού, αποχέτευση, δυνατότητα υγειονομική περίθαλψη που πλήττει τα παιδιά και να παρέχονται και άλλε υπηρεσίε και θέλουμε να καλύψουμε ε, και τη βία, την σεξουαλική και με βάση το φύλλο. Θέλουμε να υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό και ταχείε προτεραιότητε, αυτέ που αναφέρθηκαν νωρίτερα, αλλά δυστυχώ δεν έφτασαν ε, στο επίπεδο στήριξη από του δωρητών για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Καλωσορίζουμε λοιπόν την εκκίνηση της, του νέου σχεδιασμού, του σχεδίου για την ανταπόκριση στην ανθρωπιστική του ΕΡΑΚ. Θα βοηθήσουμε, ελπίζω, τι ανθρωπιστικέ οργανώσει να μαζεύουν τα χρήματα που απαιτούνται για να δώσουν απαιτούμενη βοήθεια ε, στους πληττόμενους ε, Ιρακινούς. Όπως είπα και στην αρχή, σίγουρα έχουμε ανταποκριθεί και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και στο μέλλον. Έχω μια ερώτηση, ε, διότι υποτίθεται ότι έχουμε σύστημα ερωταπαντήσεων. Θα είμαι θα ευγνώμονε για περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με το πώ η ανθρωπιστικό αυτό σχεδιασμό θα ταιριάξει με το στρατηγικό σχέδιο και τι προτεραιότητε fast track. Αυτά τα τρία, ε, τρεις στοιχές πρέπει να συντονιστούν για να έχουμε αποτελεσματική παροχή της βοηθείας. Πώς θα γίνει αυτό, αυτή είναι η ερώτησή μου και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κέλλη Κλέμενς που είναι αναπληρώτρια γραμματέας ε, του Γραφείου Μετανάστευσης ε, Πληθυσμιακών Υποθέσεων των ΗΠΑ. Ευχαριστώ εδώ στα κίτρινα, στη μέση είμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένα Έθνη που διοργάνωσαν αυτή τη σημαντική συνάντηση για να ρίξουμε το φως στο θέμα του Ιράκ και των τεραστίων ανθρωπιστικών αναγκών που υπάρχουν στη χώρα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ήμασταν έθερμον ε, έθεμε υποστηρικτή στον ευάλωτο Ιρακινό στην περιοχή και είμαστε ικανοποιημένοι που η περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν και η κυβέρνηση του Ιράκ συνεργάζονται για να εντοπιστούν οι ανάγκε των αμάχων που έχουν ξεφύγει από τι χώρε του λόγω των μαχών από την αρχή τη κρίση του Ιράκ. Η ΕΠΑ ήταν μεγάλο ε, συνέδρα με τα μάλα. Ε, ε, δώσαμε πάνω από 407 εκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια για τους εκτοπιστέντες Ιρακινούς συμπεριλαμβανομένων 208 εκατομμυρίων φέτος και μόνο και περισσότερα από αυτά ανακοινώθηκαν στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού που ήρθε στη Ουάσιγκτον. Ε, μιλήσαμε πολύ για τι ελλείψει χρηματοδοτήσεω σήμερα το πρωί και τι έκτατε ανάγκε που εξακολουθούν να ξεπερνούν τι ανθρωπιστικέ ανάγκε και τι ανταποκρίσει τη διεθνού κοινότητα Η Γκράντε και άλλοι είπαν ότι τώρα είναι η στιγμή να αντιδράσουμε διότι είναι κρίσιμη στιγμή που αντιμετωπίζουν τα προγράμματα βοηθεία στο Ιράκ και θέλουμε άμεση ανταπόκριση στι ανάγκε που έχουν περίπου 3 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπιστέντε η ανθρωπιστική ανταπόκριση θα πρέπει να δοθεί άμεσα από την κοινότητα και να προβλέψουμε και άλλους εκτοπισμούς και θα πρέπει να επενέσουμε τον μηχανισμό ταχείας ανταπόκρισης που υποστηρίξαμε μαζί με την ΕΚΟ αλλά αυτοί οι πόροι θα εξαντληθούν μέχρι το τέλος του μηνός ε, του επομένου και χρειάζεται άμεση στήριξη. Είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία και επώδυνη των διαφόρων κόμβων του ανθρωπιστικού συστήματος. Ε, για να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το πρόγραμμα το ανθρωπιστικό περίεργο Λύση το πρωί και να δώσουμε ευκαιρίε να ευχαριστήσω όλου εκείνου που ε, άοκνα εργάστηκαν προσωπικό κίνδυνο για να δώσουν τη βοήθεια στου εκτοπιστέντε Ιρακινού και άλλου που πλήττονται από τη σύγκρουση. Δοθήσει τη διαδικασία θέσεω προτεραιοτήτων που απαιτείται για να ε, σχεδιαστεί σωστά το πρόγραμμα, χρειάστηκε περιφερειακό συντονισμό. Τονίστηκε η ολιστική προσέγγιση στο Ιράκ και χαιρόμεθα γι' αυτό. Και πέρα από τις άλλες μεθόδους θέλουμε να καλυφθεί όλο το Ιράκ και το νότιο Ιράκ και το κεντρικό Ιράκ πέρα του βορείου και επικροτούμε τη συμπερίληψη μια στρατηγικής εξόδου και πώς συναρτάται αυτό με τις ευθύνες της κυβερνήσεως του Ιράκ εναντί του λαού του. Ευχαριστούμε γι' αυτό και για να πηχήσω αρκετούς ομιλητές σήμερα το πρωί η πρόσβαση προς τους εκτοπιστέντες είναι κρίσιμη προτεραιότητα για μας πρέπει να γνωρίσουμε τι ανησυχίε που υπάρχουν στην ασφάλεια, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξισορροπήσουμε του περιορισμού για την ασφάλεια και ανθρωπιστικέ αρχέ. Είναι επιτακτική ανάγκη διότι προβλέπουμε σημαντικέ μελλοντικέ ροέ εκτοπιστέντων, διότι γίνονται μάχες, ε, επεκτείνονται μάχε σε άλλε περιοχέ. Οι εκτοπιστέντε ε, δεν θα έχουν πλέον ασφαλεί περιοχέ να πάνε και όλοι οι εκτοπιστέντες ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεπιθήσεων και φιλετικής καταγωγής θα πρέπει να μπορούν να επιστρέψουν αν το θέλουν στις αιστείες τους ασφαλώς. Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε για να συζητήσουμε το θέμα σήμερα και να είμαστε εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει κι άλλοι το λόγο, αλλά ο χρόνος ε, πιέζει και θέλουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις. 10-15 λεπτά απαντήσεις ε, έχουμε με τρόπο ευέλικτο, διαδραστικό, δεν ξέρω ποιος επιθυμεί να αρχίσει. No, just Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα, λέει ο κύριος Τούρκο, να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις από την Αντιπρόεδρο Γκόμους, παραδείγματος χάρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να Ξέρουμε από πού προέρχεται αυτή η ανθρωπιστική ανταπόκριση. Ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει συνεργάζονται με ε, τους οργανισμούς του ΟΗΕ και βασίζονται σε αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν συμμετέχουν χώρε ε, τη περιοχή για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. και πρέπει να βασίζουμε τη δράση μας ε, σε βασικές αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου. Οπωσδήποτε λοιπόν θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Θα ήθελα μόνο να κάνω μια, ένα σχόλιο για την Τουρκία. 1,7 συρι πρόσφυγες ε, είναι, ένα ε, πρόσφυγες είναι στην Τουρκία και 92.000 επίσης ε, Ιρακινοί βρίσκονται στην Τουρκία και η... παρά το, τη μαζική ε, προσέλευση ε, προσφύγων έχει περάσει από το τουρκικό κοινοβούλιο μια νέα νομοθεσία για το άσυλο και έχει αναλάβει πράγματα που ε, νωρίτερα ήταν αρμοδιότητα του ΟΗΕ. Θα έπρεπε λοιπόν να το αναγνωρίσουμε αυτό διότι έχουν παρέσχει πόρους ε, για τους πρόσφυγες. Αν ε, δεν υπήρχαν αυτά θα ερχόντουσαν πολύ περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Για την σεξουαλική βία, γιατί αναφέρθηκε σε αυτό η κυρία Γκόμες, υπάρχει μια μεγάλη συνιστόσα του σχεδίου που ε, αφορά σε αυτό το θέμα και επιτόπου υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που διεξάγονται σε συνδυασμό με την κουρδική κυβέρνηση ακριβώς για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ε, των ε, κοριτσιών και των γυναικών που έχουν υποστεί αυτή την αποτρόπια σεξουαλική βία. Η τρίτη συνιστόσα και τώρα θα κάνω μάλλον και ένα γενικό σχόλιο. Πέρυσι για την επανεγκατάσταση είχαμε 80.000 περίπου ε, και από τις ευρωπαϊκές χώρες ε, το αντίστοιχο σταθμό είναι 8.500. Βλέπουμε ότι θα πρέπει η ποσόστοση να αυξηθεί σημαντικά. Είναι πολύ σημαντική η πρόταση που κατέθεσε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποσόστοση επανεγκατάστασης 20.000 ανθρώπων. Έτσι δίνεται εν μέρη μια απάντηση τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Η κυρία Νόσουόρθη. Ήθελα να απαντήσω για το τρόφιμα στα σχολεία. Στο Ιράκ, Συρία, στην περιοχή γενικότερα, στο Νότιο Σουδάν και αλλού, κινδυνεύουμε να υπάρξει μια ολόκληρη γενιά που να θεωρεί ότι η βία είναι απάντηση τι κάνουμε εμείς λοιπόν στο παγκόσμιο επιστημιστικό πρόγραμμα όταν έχουμε τα χρήματα, γιατί είναι εθελοντικές οι συνδρομές, ε, από αυτό εξαρτόμαστε. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές και την αυτοδιοίκηση και τις κυβερνήσεις για να δίνουμε μας στα σχολεία ε, και σε αγόρια και σε κορίτσια γιατί είναι σημαντικό να μεν και εκεί λοιπόν και στο Νότιο Σουδάν και στη Συρία και σε ε, μερικά από τα πιο δύσκολα και σκληρά μέρη του κόσμου το κάνουμε αυτό και συνδυάζουμε την εκπαίδευση με τη διατροφή και με άλλους οργανισμούς, με τη UNICEF, ε, είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και με άλλες οργανώσεις για να μην χάσουμε μια γενιά ολόκληρη. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό είναι μια κατάσταση που αλλάζει ραγδαία και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο. Θα ήθελα λίγο να μιλήσω και για την Τουρκία και για το σχόλιο αυτό. Η δική μας εμπειρία είναι ότι η τουρκική κυβέρνηση αποδείχθηκε πάρα πολύ γενναιόδορη στην αντιμετώπιση αυτής της επιστημιστικής ασφάλειας και τονίζω αυτό που είπε ο συνάδελφος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έγκελαντ μου ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολλά σωστά υπόθηκαν και χαίρομαι που πολλοί ομιλητές ε, ε, δώσαν έμφαση στη σημασία να δοθεί όθηση για πολιτική λύση. Διότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει να σφυριλατηθεί διάλογος. Οι περιφερειακές δυνάμεις, οι διεθνείς δυνάμεις θα πρέπει να ενωθούν αντί να διαγωνίζονται εκεί στο Ιράκ. Μπορούν οι πάντες να κάνουν περισσότερο και οι γείτονε και οι περιφερειακοί παράγοντες και οι διεθνείς. Αυτό που βλέπουμε τώρα όμως είναι ένα ντόμινο. Έχεις άλλη συνδοτή αντίδραση ε, ε, αρνητικών καταστάσεων. Ο κόσμος ε, πολλώνεται και περιθωροποιείται διότι εκτοπίζεται συνεχώς και συνεχώς υπήρχαν κάποια στοιχεία σταθερότητα και υπάρχουν ακόμα, αλλά έχουν υπονομευθεί. Ο εξτρεμισμός έχει να κερδίσει όταν οι πάντες χάνουν την ελπίδα τους. Ό,τι δεν κάνουμε τους επόμενους μήνες μπορεί να το μετανιώνουμε δεκαετίες ολόκληρες θα μπορούσαμε να δούμε πολύ χειρότερες σειράξεις και μετατοπίσεις πληθυσμών και τότε πραγματικά θα είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση. Όπως είπε και η εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, ε, λέμε ότι μας τελειώνουν τα χρήματα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των υπολείπων που συμμετέχουν στην ταχεία απόκριση. Αυτό δείχνει πόσο απεγνωσμένη είναι η κατάσταση. Αν αδρανίσουμε θα χαθεί και ελπίδα ε, και μπορεί να συμβούν τα πάντα. Και θέλω να τελειώσω λίγο με την παιδεία. Συμφωνώ με την ε, κυρία Γκόμες που μίλησε γι' αυτό για μας. Αυτό που ακούμε από εκτοπισμένου ανθρώπου και μα εκπλήσει είναι ελπίζω τουλάχιστον τα παιδιά μου να μπορέσουν να πάνε σχολείο για να μην χαθεί αυτή η γενιά. Λοιπόν, υπάρχει το σχέδιο, χρηματοδοτήστε το, βοηθήστε μας και βοηθήστε και αυτή την πολιτική διαδικασία για να ε, αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν είναι τελείως ε, απελπίδα η κατάσταση, αλλά λίγος χρονοσμένη. Ο κύριος Γιουσέφ. Δεν θέλω να επαναλάβω τις ίδιες απαντήσεις, συμφωνώ. Και δεύτερον, δεν θα μπορέσω να απαντήσω παρά μόνο στις ερωτήσεις που απευθύνονται στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Είναι ιδιαίτερα ε, μακροχρόνια η διαμάχη στο Ιράκ δεν χρονολογείται μόνο από 18 μήνες και ό,τι και να κάνουμε σήμερα εμείς οι διεθνείς ε, οργανώσεις, τι κάνουμε, βάζουμε ένα χανζαπλάστ πάνω στην πληγή. Πρέπει να τονίσουμε πόσο μακροχρόνια είναι η σύραξη αυτή. Έχουμε εδώ πέρα ανθρώπους που έχουν ε, ζήσει την σύραξη από την αρχή και μπορούν να μας τα πούνε. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κουμιουαχάν που είναι αναπληρώτρια γραμματέας για ανθρωπιστικά ζητήματα και για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ε, του πάνελ και του ακροατήριο. Είναι πολύ εύστοχα τα σχόλιά σας. Νομίζω η πρέσβη από τον Καναδά ε, μου έκανε μία ερώτηση για την επιχείρηση που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Πρόκειται, ναι, για μία νέα προσέγγιση. Έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ η κατάσταση και αυτή είναι η απάντηση που δίνουμε επί σας είπα, είναι μια μινιμαλιστική ευσταμένη προσέγγιση για τα απολύτως χρειαζόμενα. Μετά το πρώτο εξάμεινο θα προκύψει νέο ε, σχέδιο έκτακτες ανάγκης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση της ε, σημερινής ε, εκδήλωσης και όλοι οι προσκεκλημένοι μπορούν να τραβήξουμε την προσοχή σε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Ιράκ. Μιλήσατε όλοι για τα βάσανα του Ιρακινού λαού και αυτοί που αγωνίζονται επί τόπου, η Λις Γκράντε που τους καθοδηγεί έχει ε, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ε, καταφέρει να κινητοποιήσει μέσα από αυτόν τον μηχανισμό που ανέφερε επανειλημμένα να φτάσει η βοήθεια σε αυτούς που δεν χρειάζονται περισσότερα και ε, νομίζω ότι αυτό το response plan, το νέο σχέδιο είναι Ό,τι καλύτερο έχω δει προκύπτει ε, από τις προσπάθειες που γίνονται επί τόπου και η Λις Γκραντ το περιέγραψε με εξαιρετική ακρίβεια οι βασικές αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου για τις ενόπλες σειράξεις, η βασική ε, αξιοπρέπεια παραβιάζονται καθημερινά και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την προστασία που πρέπει να προσφέρουμε και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία το θέμα της προστασίας στο νέο σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Στο μεταξύ όμως έχουμε καθήκον για αυτούς που εξακολουθούν να έχουν ελπίδα, όπως είπε κάποιος από το ε, πάνελ, την ελπίδα ότι κάποιος θα έρθει να τους προστατεύσει. Και Τόνι το είπες και εσύ, έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτή ακριβώς την ελπίδα που έχουν παρά το ότι θα αντιμετωπίσουμε ακόμη μεγαλύτερες ε, δυσκολίες προσεχεί μήνες. Ε, απευθύνουμε θερμή, θερμή, θερμότατη έκκληση προς τους πολιτικούς και του εμπλεκόμενους φορείς ε, να μας βοηθήσουν με τη χρηματοδότηση ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε αυτούς που μας χρειάζονται τώρα για να σταματήσουν τα βάσανά τους να σταματήσει αυτή η ανθρώπινη τραγωδία, αυτή η καταστροφή. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο και την ε, Γενική Διεθνή ΕΚΟ. Σίγουρα θα μεταφέρουμε αυτό το ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης προς τον Ιρακινό λαό. Ευχαριστώ πολύ. Για να κλείσουμε. Ε, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Στυλιανίδη που είναι Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Ελπίζω να ακούσατε όλα αυτά που υπόθηκαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξοχότητες, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Απειρωτή Γενικό Γραμματέα και όλους τους ε, ομιλητές της εκδήλωσης μας δόθηκε μια γενική εικόνα όσον αφορά τις ανθρωπιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στο Ιράκ. Παρουσιάσατε τα βασικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για ισχυρότερη ανθρωπιστική προσπάθεια, προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας, συμμετοχή αυτής. Όπως ακούσαμε από τη Λίζα Γκράντε, το νέο σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράκ δείχνει ξεκάθαρα ότι χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια μέχρι το τέλος του έτους. Ο Άντωνι Λέικ αναφέρθηκε στα δεινά που περνούν τα παιδιά. Η κυβέρνηση του Ιράκ και η περιφερική κυβέρνηση του Κουρδιστάν αντιμετωπίζουν μεγάλη πρόκληση. Να συντηρούν τις προσπάθειές τους, να συντηρούν το συντονισμό που απαιτείται για να εξασφαλίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια. να παρέχονται βασικές υπηρεσίες στους πληγέντες πληθυσμούς. Πάντα ανεξάρτητα της θρησκείας την οποία ανήκουν ή της κοινότητας ή της ταυτότητας των ανθρώπων. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να εγκαταλείψει τα θύματα της σύγκρουσης στο Ιράκ, των συγκρούσεων στο Ιράκ. Πρέπει τώρα να δράσουμε, όχι αύριο. Όπως είπα και κατά τη διάρκεια της παρέμβασης μου, της αρχικής, θα πρέπει να εγγυηθούμε την ασφαλή ανθρωπιστική πρόσβαση άνευ όρων. Σημαντικότατο, δυσχερέστατο. Το ξέρεις καλύτερα από μένα, Λίζ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την παροχή της βοήθειας. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε εκείνους που έχουν ανάγκη. Άνευ διακρίσεων. η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται βάσει των ανθρωπιστικών αρχών, βάσει των αναγκών. Όλα τα εμπλεκόμενα σύραξη μέρη πρέπει να ε, συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει ε, διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να σεβαστούν και να προστατεύσουν όλους τους άμαχους. Τώρα όσον αφορά την κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών θα πω ότι είναι ηθική υποχρέωση. Αυτό το αναφέρατε πολλοί από εσά. Είναι επιτακτική ηθική ανάγκη. Πέραν αυτού είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια και την σταθερότητα. Όχι μόνο για την χώρα αλλά για όλη την περιοχή. Ίσως και για όλο τον κόσμο είναι σημαντικό αυτό, για την ασφάλεια όλου του κόσμου. Εάν δεν καλύψουν αυτές τις ανάγκες, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε έφορο έδαφος για περαιτέρω συγκρούσεις. Οι άμαχοι τελικά θα είναι θύματα ε, τρομοκρατικών οργανώσεων όπως είναι το Ισλαμικό κράτος. Ο φαύλος κύκλος της βίας θα συνεχιστεί. Αγαπητοί φίλοι, η λιλεγγύη της Ευρώπης προς το Ιράκ είναι στέρεη, είναι απτή. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα μεταφέρω στην αποστολή μου στο λαό του Ιράκ. Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις μας. Πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέσα Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη, είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής για τα ανθρωπιστικά θέματα στο Ιράκ. Μέχρι τώρα, φέτος, έχουμε διαθέσει πάνω από 38 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική χρηματοδότηση. Η κλιμάκωση των μαχών ασκεί περαιτέρω πιέσεις στους περιορισμένους ανθρωπιστικούς πόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ανταπόκριση σε αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεθάρρυνε τους εταίρους της να εξασφαλίσουν την παροχή βασικής βοηθείας. Δηλαδή νερό, τρόφιμα, αποχέτευση, ε, αντικείμενα υγιεινής, κυρίως σε τομείς που έχουμε τις περισσότερους εκτοπιστέντες. Είμαι υπερήφανος που σας λέω σήμερα ότι ανακοίνωσα άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστικής βοηθείας ότι θα διατεθούν. Αυτό είναι το ποσό που μπορώ να διαθέσω τώρα. Θέλω να είμαι σαφής. Έχουμε μακροπρόθεσμη δέσμευση που έχουμε αναλάβει. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες όσο υπάρχουν ανάγκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθεί να είναι στην πρώτη γραμμή της κάλυψης των αναγκών, όσο και αν χρειαστεί. Όχι μόνο οικονομικής ενίσχυσης, αλλά θα προωθούμε τον σεβασμό των διεθνών ανθρωπιστικών αρχών και του διεθνούς δικαίου, προωθώντας πολιτικές λύσεις. Για αυτό το σκοπό όμως θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συνεργαστούμε. Χρειαζόμαστε συλλογική υποστήριξη διότι και η ευθύνη είναι εκείνη. Και οι δράσεις μας πρέπει να είναι κοινέ. Μόνο ότι ούτω τρόπος θα μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά, την πραγματική διαφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες ε, και όσους μίλησαν. Ας ελπίσουμε ότι η σημερινή συνεδρίαση θα ε, βοηθήσει και θα είναι μια κραυγή ευθύνης και αγωνίας ε, και ε, όχι μόνο εμείς αλλά και οι διάφορες οργανώσεις βοηθούν. Αυτά. Επόμενες συνεδριάσεις ΔΕΒΕ 15-16 Ιουνίου στις Βρυξέλλες και ΑΦΕΤ 11 Ιουνίου στο Στρασβούργο λήξη συνεδρίασης.